Κυρίε Κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω όλους. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας, την πρώτη μας συνεδρίαση. Και σήμερα το απόγευμα μπορούμε να καλωσορίσουμε την Υπουργό Υπηρεσιμών και Ανωτέρα Εκπαίδευση τη Πολωνία, που ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυρία Μπάρμπαρα Κουντρίτσκα, πρώην συναδελφό μας και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία σας καλωσορίσω στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας εδώ, χαιρόμαστε για αυτά τα οποία θα μας αναφέρετε και χαιρόμαστε φυσικά και για την Πολωνική Προεδρία. Σας ευχαριστώ λοιπόν και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν δουλεύει αυτό το μαραφέτη. Όχι πραγματικά. Oh, Εντάξει, λειτουργεί τώρα. Νέε τεχνολογίε. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, τεράστιες προκλήσεις που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαμε ξανά. Γνωρίζουμε επίσης ότι βρισκόμαστε στα μέσα μιας πολύ σοβαρής κρίσης, χρηματοπιστωτικής κρίσης καταρχήν και υπάρχει όλο και λιγότερη εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ένας από τους στόχους λοιπόν της Πολωνικής Προεδρίας είναι να βάλει ένα τέλος στην κρίση. Δεν είναι όμως αυτός ο μόνος μας ε, στόχος. Άλλος ε, στόχος μας είναι να επιστρέψουμε σε μια γρήγορη οικονομική ανάπτυξη. Είμαι πεπισμένη ότι η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας αποτελεί ένα στοιχείο κλειδί το οποίο θα μας βοηθήσει να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον σε όλους τους πολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πετύχουμε όμως αυτό το στόχο, την οικονομική δηλαδή ανάπτυξη, μέσω ευφυών δραστηριοτήτων, αυτό θα μπορέσουμε να το πετύχουμε μόνο εφόσον χρησιμοποιήσουμε πλήρως όλες τις κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες που έχουμε. Και τέτοιες ευκαιρίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες μέλη, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα μάλιστα πρέπει να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως το κεφάλαιο διανόησης που διαθέτουμε εδώ στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια κοινότητα σοφίας, ταλέντου, γνώσης. Η γνώση και η εμπιστοσύνη είναι τα στοιχεία που χρειάζονται για να προχωρήσουμε. Είναι αυτά τα οποία θα επιτρέψουν σε όλο τον κόσμο να προχωρήσει. Η Πολωνία λοιπόν είναι η χώρα εκείνη η οποία κατάφερε να αποτελέσει έναν πράσινο θύλακα ανάμεσα στις χώρες οι οποίες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Και αυτό γιατί η Πολωνία κατάφερε όχι να ξεπεράσει την κρίση, αλλά είναι μια χώρα όμως η οποία βασίζεται στους νέους, στο ταλέντο τους, στις ικανότητές τους. Πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε. Έτσι λοιπόν πιστεύουμε στην Πολωνία ότι αυτό το κεφάλαιο ε, γκρίζα ουσίας που διαθέτουμε πρέπει να αποτελέσει και την προτεραιότητα για την Πολωνική Προεδρία. Η ίδια βέβαια η Προεδρία από μόνη της δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα και να διακανονίσει τα πάντα. Χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων και όλος ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειαζόμαστε επίσης συνεργασία με τις χώρες μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να πετύχουμε τους κύριους στόχους μας. Συγχρόνως όμως θα συνεργαζόμαστε και με την Δανέζικη Προεδρία και με τους Κύπριους συναδέλφους που θα αναλάβουν μετά, προκειμένου το πρόγραμμά μας να είναι κοινό, να είναι το πρόγραμμα του τρίου της ε, τριμερούς αυτής ε, προεδρίας και να πετύχουμε τους στόχους μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βγει πιο ισχυρή από την κρίση εφόσον μπορέσει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της. Η στρατηγική για την Ευρώπη 2020 πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή αποτελεσματικά από τα κράτη-μέλη και από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα επικεντρωθούμε σε μια ανάπτυξη που να είναι βιώσιμη, στην οποία να συμπεριλαμβάνονται όλοι. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προωθήσει νέες πηγές ανάπτυξης, όπως είναι το κεφάλαιο αυτό, η γκρίζα ουσία, όπως επίσης και μια πολιτική που να βασίζεται στην οικονομία της γνώσης. Θα αντιμετωπίσουμε έτσι τις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις και ότι προκλήσεις υπάρχουν σχετικά με το περιβάλλον, την ε, τον ασφαλή εφοδιασμό ενέργειας και την βιοπικιλότητα. Μελλοντικέ οικονομικές επιτυχίες δεν θα είναι εφικτές παρά μόνο αν αυξήσουμε τις επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει για να πετύχει και να εφαρμόσει το τρίγωνο της γνώσης, έτσι ώστε να έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό χώρο έρευνας που θα μας επιτρέψει να μην έχουμε κατακερματισμένες πολιτικές και να έχουμε πραγματικά κέντρα ερευνητών. Μια τέτοια στρατηγική μπορεί να βοηθήσει και την καινοτομία και να ε, βοηθήσει να έχουμε τα βέλτιστα δυνατόν αποτελέσματα από την έρευνα και την καινοτομία χρησιμοποιώντας περισσότερο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στην διαδικασία καινοτομία και στηρίζοντας επίσης και πλήρως την γκρίζα ουσία της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά σε αυτά τα πλαίσια. Γνωρίζουμε όλοι την διαδικασία για να πετύχουμε τους στόχους μας, ότι η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει και μάλιστα όχι μόνο εγκρίνοντας τη νέα στρατηγική που ονομάζεται Ευρώπη 2020, αλλά επίσης υιοθετώντα και εμβληματικές πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες υπέρ της καινοτομίας για παράδειγμα, που είναι μια από τις πιο σημαντικές εμβληματικές πρωτοβουλίες. Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα τον Νοέμβριο που μας πέρασε υιοθέτησε συμπεράσματα και τα συμπεράσματα αυτά αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό βήμα και μια συνεισφορά στην συζήτηση που ξεκίνησε και γίνεται στο Συμβούλιο για την Καινοτομία. Η Πολωνική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή τέτοιων πρωτοβουλειών και λύσεων που απορρέουν από την εμβληματική αυτή πρωτοβουλία υπέρ της καινοτομίας. Χρειάζονται επίση επενδύσει στον τομέα τη έρευνα, τη κατάρτιση, τη εκπαίδευση και τη καινοτομία βέβαια. Πράγματα στοιχειώδη που αποτελούν και το άνισμα για να οδηγηθούμε στην ανάπτυξη. Τέτοιε δραστηριότητε μα βοηθούν να δημιουργήσουμε καλέ οικονομικέ προποθέσει από τη μία και από την άλλη θα είμαστε και σε θέση να αντιδράσουμε απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις του πολιτισμού μας. Έτσι θα μπορέσουμε επίσης όλες αυτές τι δραστηριότητες να τις ε, χρησιμοποιήσουμε για την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Αυτό στο κάτω-κάτω είναι και ο στόχος της στρατηγικής 2020. Στρατηγική, η οποία βέβαια έχει και άλλους στόχους, όπως για παράδειγμα το 2020 να έχουμε πετύχει 3% των δημοσίων δαπανών της κάθε χώρας που να πηγαίνει στην έρευνα και η χρηματοδότηση αυτή να μην γίνεται μόνο από το δημόσιο αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να ξεχνάει τα θεμέλια της, τις βάσεις της. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι υπεύθυνη όχι μόνο και να λογοδοτεί, όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά της όργανα, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε και να οδηγηθούμε σε τέτοιες αλλαγές και τροποποίησεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ώστε να μπορούμε στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό της Ευρώπης που προέρχεται από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε εξαίρετη, τους ερευνητές, πρέπει λοιπόν να τους χρησιμοποιήσουμε και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε ήδη στην αρχή της διαδικασίας αυτής να ξέρουμε ότι όλοι είναι ίσοι και ότι όλοι έχουν εξίσου πρόσβαση στη διαδικασία αυτή. Να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και την έρευνα και την καινοτομία ε, προς όφελος των περιοχών που βρίσκονται πιο πίσω. Ορισμένες χώρες μέλη και ορισμένες περιφέρειες όντως δεν εκπροσωπούνται παρκώς στις προτεραιότητες αυτές. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Για να γίνει αυτό πρέπει να θυμόμαστε και να χρησιμοποιούμε ε, μέτρα σύγκρισης για να μπορούμε να μετρήσουμε την ανάπτυξη. Το Συμβούλιο λοιπόν προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης, βαθμολόγησης. Έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε την πρόοδο που επιτυχάνεται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας στις διάφορες περιφέρειες και χώρες της Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις σημαντικές προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια και ότι τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας Πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε με συνοχή να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και με κοινέ δράσεις. Και όταν λέω κοινέ δράσεις, ενώ ότι πρέπει να υπάρχει συντονισμός μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των χωρών μελών. Άρα χρειάζονται κοινέ ε, πρωτοβουλίες και κοινό προγραμματισμός. Χρειάζεται μια εταιρική σχέση υπέρ της καινοτομίας με πειραματικά προγράμματα. Η Ευρώπη χρειάζεται έναν κοινό χώρο έρευνας για να ενθαρρύνει τα καλύτερα ταλέντα και χρειάζεται και μεγάλες επενδύσεις. Αυτές πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη. Η διαδικασία ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας θα ολοκληρωθεί το 2014. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την κοινή αγορά για την έρευνα, την καινοτομία και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε θα αναπτυχθούν ώστε να είναι έτοιμα εν ώψη των νέων δημοσιονομικών προπτικών. Είναι ζωτική σημασία να φροντίσουμε να υπάρχει κινητικότητα μεταξύ των ερευνητών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να είναι αυτοί ικανοί να χρησιμοποιούν τις υποδομές για την έρευνα που υπάρχουν. Όλοι οι επιστήμονες, όλοι οι ερευνητές πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση στις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι οι δραστηριότητε αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Προεδρία θα πάνε προ αυτή την κατεύθυνση. Θα προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα συντονίσουμε με την ατζέντα και τη Κομισιόν και του Συμβουλίου. Οι δραστηριότητε μα, λοιπόν, αυτό το εξάμεινο, αυτέ θα είναι για να ενισχύσουμε το πρόγραμμά μας που ονομάζεται Horizon. Horizon. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πλαίσιο, ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο πρέπει να είναι πιο φιλικό, πιο απλό και προς όφελος ακόμα περισσότερο υπέρ των χρηστών του. Ειλικρινά, επιθυμούμε να έχουμε ε, ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα χάρη στο συντονισμό μεταξύ μας και χάρη της συνοχής. Χάρη των, του Ταμείου Συνοχής που είναι στη διάθεση των χωρών μελών. Θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες. Και όταν λέω διαδικασίες εδώ, εννοώ τις διαδικασίες χρηματοδότησης, και τις διαδικασίες εξέβρεσης χρηματοδότησης για τα διάφορα προγράμματα. Εδώ θέλω να υπάρξει απλοποίηση. Απλοποίηση όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα και απλοποίηση επίσης για όλα τα μέσα που έχουν να κάνουν με διοικητικά ζητήματα. Η συζήτηση αυτή θα λάβει χώρα όχι μόνο στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν θα συζητήσουμε για το μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο, Ελπίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει στα τέλη Νοεμβρίου έτοιμο ένα πρώτο σχέδιο. Επιπλέον θέλουμε να οργανώσουμε και διάφορες διασκέψεις, μια ευρεία διαβούλευση καλύτερα, διαβούλευση για τις ιδέες που παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο είναι μια διαβούλευση που έχει αναγγείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμείς στην Πολωνία θα οργανώσουμε μια ενδιαφέρουσα νομίζω συνδιάσκεψη η οποία θα λάβει χώρα 19 και 20 Οκτωβρίου. Στην διάσκεψη αυτή θα συζητήσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με ένα νέο νομοθετικό πακέτο το οποίο θα αποτελεί μέρος του νέου προγράμματος πλαισίου. Είμαστε λοιπόν ευγνώμονες και το λέμε αυτό για την ε, ε, Ουγγρική Προεδρία. Το γύρο βάτων που ξεκίνησε ήταν κάτι πολύ σημαντικό και ελπίζουμε και εμείς να μπορέσουμε να βρούμε τεχνικές λύσεις σε ό,τι δυσκολίες υπήρχαν, όπως επίσης και ένα κανονισμό. Περιμένουμε πάντως τα συμπεράσματα από ένα πειραματικό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εταιρικής Σχέσης όσον αφορά την γύρανση του πληθυσμού. Πληθυσμός που γερνάει εν υγεία. Όλα αυτά θα συζητηθούν σε συνεδρίες του Συμβουλίου που θα γίνει στις Βρυξέλλες. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για διάφορες εταιρικέ σχέσεις που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και για διάφορα κοινά προγράμματα, παρά τις όποιες διαφορές έχουμε μεταξύ μας. Και αυτό γιατί τα διάφορα ιδρύματα τεχνολογίες έρευνας και τα λοιπά έχουν κοινά, έχουν και διαφορές μεταξύ τους. Καλό είναι λοιπόν μεταξύ τους να μπορούν να συνεργαστούν βασιζόμενοι στα κοινά 10 και 11 τώρα του μηνό στην ε, Βαρσοβία οργανώνουμε την τρίτη διάσκεψη κορυφής για την καινοτομία. Στη διάσκεψη αυτή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα. Αυτό που είναι επίσης πολύ σημαντικό προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο την κρίζα ουσία που διαθέτουμε στην Ευρώπη, να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχει ήδη στη διάθεσή της η Ευρώπη να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή πιο αποτελεσματικά τα, από τα πανεπιστήμια, την καινοτομία και την έρευνα. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα κατά την πρώτη υπουργική διάσκεψη που θα προηγηθεί ενός συμβουλίου που θα λάβει η χώρα στο Σόμποτ στις 20 Ιουλίου, πολύ σύντομα δηλαδή. Επιπλέον, Υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες που προγραμματίζουμε. Για παράδειγμα, όσοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Marie Curie θα βρεθούν μαζί στα πλαίσια μιας διάσκεψης στην Κρακοβία που θα οργανώσουμε και θα αποτελεί μέρος του Atomium Culture. Όλα αυτά τα γεγονότα, όλες αυτές οι εκδηλώσεις θα μας επιτρέψουν να συζητήσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να τις θυμόμαστε τις προκλήσεις αυτές όταν ετοιμάζουμε το νέο πρόγραμμα πλαίσιο και ε, καθορίσουμε τις αρχές του. Η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται και σε πολιτικό και σε επιστημονικό επίπεδο και σε πολιτικούς και σε επιστημονικούς κύκλους. Και εσείς βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχετε στη διαβούλευση αυτή. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα μαζί για το μέλλον της ευρωπαϊκής καινοτομίας. Καινοτομία η οποία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα για να πετύχουμε την οικονομική ανάπτυξη. Ιδιαίτερα σήμερα που περνάει από τόσες δυσκολίες η Ευρώπη. Η καινοτομία είναι μία από τις πιο βασικές λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι κάτι που δεν το διαπραγματευόμαστε, δεν νομίζω ότι είναι ένα επίμαχο θέμα. Συμφωνούμε όλοι από αυτού ότι η καινοτομία δηλαδή είναι ένα από τα βασικότερα κεφάλαια που έχουμε στη διάθεσή μας. Από εδώ και πέρα να ακούσω τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας για ό,τι θέμα θέλετε να θίξετε. Ό,τι θέλετε θα σας ακούσω ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Νομίζω ότι από αυτά που ακούσαμε είναι σαφές ότι το μέλλον της Ευρώπης <clears throat> εξαρτάται από το αν θα μπορέσουμε στον τομέα της ε, έρευνας και της καινοτομίας να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Επομένως δεν αρκούν μονάχα τα λόγια, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε πράγματι αυτούς τους στόχους. Ο κύριος Γκίρεκ είναι ο πρώτος ο οποίος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Καλό απόγευμα σε όλου. Θα ήθελα να καλωσορίσω ε, την Υπουργό, να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είσαστε και πρώην συνάδελφο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και μια επιφανής νομικό στη χώρα μα. Και χαιρόμαστε που μα παρουσιάζετε θέματα όπω οι επιστήμες και η έρευνα, διότι οι επιστήμε είναι η βάση τη καινοτομία και η καινοτομία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην αγορά και στην, στην αγορά και η καινοτομία θα μας επιτρέψει ε, ε να είμαστε ανταγωνιστικοί από αυτήν εξαρτάται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα πριν, πριν σχολιάσω αυτό το θέμα να πω ότι υπάρχει κάτι το οποίο επηρεάζει την όλη πολιτική καινοτομία. Εδώ είμαστε στην Επιτροπή Ήτρε, δηλαδή μια επιτροπή που ασχολείται με τη βιομηχανία, με την έρευνα, την επιστημονική έρευνα ε, και με επιστημονικά θέματα εν γέννη. Και υπάρχει κάτι το οποίο φαίνεται ότι κυριαρχεί στις δραστηριότητές μας σε αυτήν εδώ την Επιτροπή. Και πιστεύω ότι υπάρχει ένα λάθος. Μας έβαλε σε πειρασμό αυτό το δόγμα, αν θέλετε, αυτή η ιδέα. Όμως που μας οδήγησε και σε κάποιες πρωτοβουλίες, πρωτοβουλίες πολύ σημαντικές. Αλλά το πρόβλημά μου ποιο είναι, το δόγμα αυτό είναι αληθινό ή όχι. Τι εννοώ και ίσως κάποιους τους εκπλήξω. Λέγεται ότι το διοξίδιο του άνθρακα επηρεάζει την, το κλίμα. Τα διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας, θα γίνει μία σύνοδος στον Ταρφούρ για την, ε, της για τις κλιματικές αλλαγές. Βέβαια υπάρχουν και άλλες συναντήσεις, αλλά κάθε φορά οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχαναν αν θέλετε στον, στον διάλογο και αυτό για πολλούς λόγους. Αλλά ένας από τους λόγους ήταν ότι... Ε, ε, ένας από τους λόγους που έχαναν ε, σε αυτή τη συνάντηση στο Ντάρμπαν ήταν ότι έλεγαν πρέπει να σταματήσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα τελεία. Δεν προχωρούσαν περαιτέρω. Υπάρχει ένα πάνελ για, την, για τις κλιματικές αλλογές που ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις επιπτώσεις του διεξιδίου του άνθρακα. Δεν είναι όμως μόνο το διεξίδιο του άνθρακα. Υπάρχουν και άλλοι, εκατοντάδες άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν ε, το, το κλίμα. Άρα η βάση που χρησιμοποιεί αυτό το πάνελ είναι λανθασμένη. Επομένως, η πρόταση που θέλω να κάνω, κυρία Επομένως, κυρία Πρόεδρε, Ρωτώ, κυρία Υπουργέ, συγγνώμη, ρωτώ, μήπως θα πρέπει να έχουμε ένα δικό μας πάνελ, ένα ευρωπαϊκό πάνελ που να ασχολείται με τις κλιματικές αλλαγές, που θα λαμβάνει υπόψη πολλές παραμέτρους. Γιατί αυτό το ευρωπαϊκό πάνελ θα πρέπει να ε, βρει ε, τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές του κλίματος, όλες τις παραμέτρους και νομίζω ότι θα πρέπει η στάση μας να αλλάξει όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές. Διότι αλλιώς θα επηρεαστεί και η έρευνα και η οικονομία μας και η πολιτική ενεργειακή και ολοκληρώνω εδώ, Πρόεδρε, ένα παράδειγμα να σας αναφέρω μόνο. Η καινοτομία μπορεί να μας βοηθήσει να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Η καινοτομία όμως μπορεί να μας βοηθήσει ακόμα καλύτερα όσον αφορά τις, τον επηρεασμό στις κλιματικές αλλαγές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ. Έχω να θέσω το εξή ερώτημα. Εμείς εργαζόμαστε ήδη αρκετό χρόνο για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσα στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου για την επιστημονική έρευνα. Λοιπόν, τρία ερωτήματα και όχι ένα έχω, αλλά πάρα πολύ σύντομα. Θέλουμε λοιπόν κύριε Υπουργέ, να κύριε Υπουργέ, να υπάρξει μια απλοποίηση των προγραμμάτων που άπτονται της έρευνας και της καινοτομίας. Αλλά δεν είναι μονάχα μια απλοποίηση στα δημοσιονομικά. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που πρέπει να τύχουν απλοποίησης ή όχι. Δεύτερον, θα πρέπει να διατηρήσουμε μια συνέργεια των δημοσιονομικών ε, των ε, κονδυλίων με τα διορθωτικά ταμεία σε αυτό το πλαίσιο το επόμενο. Και τρίτο ερώτημα. Θα ήταν λογικό να καταλήξουμε σε μια συνεκτική κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την επιστημονική έρευνα για να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο και τι είδου δομέ θα πρέπει να εδρεώσουμε για να το πετύχουμε αυτό. Η κυρία Καρβάλιου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό και να την ευχαριστήσω για την παρουσίαση που μας έκανε. την παρουσίαση για το πρόγραμμα της Προεδρίας για την, τις επιστήμες και την Ιδιωτομία. Ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς για την απλούστευση. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η απλούστευση συμπεριλαμβάνεται στην ε, ημερήσια διάταξή σας και το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της απλούστευσης και παρακολουθεί από κοντά την εφαρμογή αυτών των μέτρων, γιατί πιστεύουμε ότι η Κομισιόν χρειάζεται πολιτική υποστήριξη για να μπορέσει να εφαρμόσει τα μέτρα απλούστευσης. Δεν είναι απλό πράγμα να, εφαρμόσει, να εφαρμόσει την απλούστευση και από τις 71 συστάσεις ε, της ε, έκθεσης ε, η Κομισιό έχει ήδη εφαρμόσει τρία, έχουμε και άλλες 40 που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση του κυρίου Όντι για την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση και μετά υπάρχουν και κάποιες άλλες συστάσεις όπου απαιτείται αλλαγή του χρηματοδοτικού κανονισμού. Πάντως προχωράμε, προχωράμε και χαίρομαι ε, και ότι υπάρχει, για το ότι υπάρχει και αυτή η ανεπίσημη, η άτυπη ε, ομάδα στο Συμβούλιο που ασχολείται με τα θέματα αυτά. Τώρα η ερώτησή μου αφορά τον προπολογισμό. Στο Κοινοβούλιο έχουμε ψηφίσει μία πρόταση που διπλασιάζει την χρηματοδότηση για το επόμενο πρόγραμμα καινοτομίας και έρευνας ε, το 7ο είναι 50, το διπλασιάζουμε. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν της 29ης Ιουνίου για τον προϋπολογισμό της κοινότητας όπου, προ, όπου προτείνονται 80 δισεκατομμύρια. Ξέρουμε δηλαδή ότι υπάρχουν και κάποια κρατημέλη τα οποία θέλουν να υπάρξει κάποια αύξηση, κάποια άλλα δεν θέλουν ε, να είναι τόσο φιλόδοξος ο κοινοτικό προπολογισμό. Εγώ θα ήθελα να ξέρω εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις και ποιες είναι οι... πώς μπορούμε να να συνεργαστούμε αν θέλετε με, τους, ε, με τα διαρθρωτικά ταμεία διότι τα, ε, έχουμε 60 δισεκατομμύρια από τα διαρθρωτικά ταμεία για την έρευνα και την καινοτομία όμως έχουμε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό ε, απορροφη, απορρόφησης των πόρων αυτών. Επομένως ήθελα να ξέρω πώς μπορούμε να απορροφήσουμε αυτά τα κονδύλια όσον αφορά τη δημιουργία του δυναμικού, να γίνει δηλαδή ε, στην αρχή της όλης διαδικασίας ε, η χρηματοδότηση. Επαναλαμβάνω, πώς βλέπετε εσείς να συνεργάζονται τα δύο ταμεία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σας παρακαλώ και πάλι να περιοριστείτε σε ένα με δύο λεπτά για κάθε ερώτημα, γιατί η κυρία Υπουργό δεν μπορεί να παραμείνει εδώ στο Δινικέ. Κύριε Οντί. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Υπουργέ για την επίσκεψή σας. Τρεις ερωτήσεις για την αναθεώρηση, τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, αξιολόγηση μάλλον του προγράμματος πλαίσιο. Έχουμε 30 δισεκατομμύρια για να δαπανίσουμε. Ε, η προκήρυξη των, δια, των, διαγωνισμών, των project, ε, για την υποβολή των project ε, έτσι όπως έχει γίνει θεωρείται ότι ικανοποιεί το, τα συμφέροντά μας έτσι όπως τα έχουμε διαμορφώσει. Και δεύτερη ερώτηση για την αναθεώρηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Στις διαπραγματεύσεις εσείς πώς βλέπετε τα κράτη-μέλη να ε, όσον αφορά τον περαιτέρω εξευρωπαϊσμό των, ε, της έρευνας. Και τρίτη ερώτηση για το Ευρατόμ. Θέλουμε να ε, προσαρμόσουμε τη διάρκεια της Ερατόμ των project Ερατόμ με, τα, με, τη διάρκεια των project των υπολείπων και ήθελα να ξέρω εσείς από πλευράς ε, του Συμβουλίου πώς βλέπετε να διαμορφώνει το θέμα αυτό. Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι δεν γνωρίζετε ενδεχομένω ότι είστε, μάλλον δεν οι συνάδελφοι, ότι είσαστε οι επικεφαλής, υπήρξατε οι επικεφαλής της καλύτερες μεταρρύθμισης που έχει κάνει ποτέ η πολωνική κυβέρνηση για τα ανθρακοριχεία και τους ανθρακορύχους Αλλά αυτό τώρα ήταν περιθωριακά μόναχα. Θέλω να έρθω τώρα σε ένα ερώτημα το οποίο αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο. Η αρχή της αριστείας λοιπόν είναι η σημαντικότερη. Είναι το στοιχείο λοιπόν κλειδί στα προγράμματα αυτά η αριστεία. Και αν ναι, με ποιο τρόπο θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η αξία και να προωθήσει και την ικανότητα καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Τι θα μπορέσει να γίνει λοιπόν σε σχέση με τα νέα κράτη-μέλη, τα οποία προς το παρόν δεν έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τα κονδύλια για την έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορέσουν λοιπόν να συμμετάσχουν στα κονδύλια αυτά. Μόνο η αριστεία λοιπόν αυτή καθεαυτή νομίζω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολύ τα νέα κράτη. Ο κύριος, η κυρία Σίζελη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Έχω τρία ερωτήματα να σας θέσω και ξεκινώ με το ερώτημα το οποίο μόλις αναφέρθηκε προηγουμένως. Είπατε ότι θα καταβάλλετε προσπάθειες να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους σε όλη την Ευρώπη. Είπατε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει και κάποια διαδικασία βαθμονόμησης, benchmarking, Και επίσης αναφέρατε ότι το δυναμικό, το επιστημονικό και το καινοτομικό που βρίσκεται στα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκμεταλλευτεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θετικό, είναι σημαντικό να μην περιοριστείτε μονάχα στα υπάρχοντα κέντρα τα οποία υπάρχουν τα κέντρα αριστείας, αλλά να δώσετε και βάση στη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξη του δυναμικού που υπάρχει. Αυτό τουλάχιστον κατάλαβα από τους λόγους σας. Δεύτερον, μιλήσατε για, τα ταμεία, για το Ταμείο Συνοχής και τη σύνδεσή του με την ε, έρευνα. Μήπως λοιπόν θα μπορούσαν τα Ταμεία Συνοχής να ευνοήσουν τα επιστημονικά ιδρύματα με προγράμματα τα οποία έχουν σε στόχο την έρευνα και την καινοτομία και πώς ακριβώς θα λειτουργήσει εδώ η συνέργεια μεταξύ τους. Επίσης, Ξέρω ότι στην Πολωνία έχετε δώσει πάρα πολύ από το χρόνο σας και την προσοχή σας στα θέματα των νέων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά σήμερα αυξάνεται η ανεργία των νέων και πάρα πολλοί νέοι βλέπουν να υπάρχει έλλειψη προοπτικών. <clears throat> Πώς βλέπετε λοιπόν αυτό το θέμα, όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά ευρύτερα. Πώς θα δώσετε προοπτική στους νέους σε όλη την Ευρώπη, αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ να σας καλωσορίσω εδώ στην Επιτροπή μας. Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας είναι το μόνο που μπορεί σήμερα να μας οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι ερευνητικές μονάδες κάνουν ό,τι μπορούν για να προσφέρουν καινοτομία προς όφελος και της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ όμως αυστηρά κριτήρια στην Ευρώπη πολύ φιλόδοξους στόχους συγχρόνως και έχουμε και διαφυγή εγκεφάλων από την Ευρώπη. Η έρευνα είτε συγχρηματοδοτείται από τη βιομηχανία, είτε οι ερευνητικές αυτές μονάδες δουλεύουν αποκλειστικά και μόνο για τη βιομηχανία. Οπότε φοβάμαι ότι τελικά οι ερευνητές ή που θα ακολουθήσουν τη βιομηχανία και η έρευνά μας θα στραφεί προς τη βιομηχανία και μόνο ή που δεν θα υπάρχει πια. Η κυρία Τόιπ. Ευχαριστώ. Μία... Η παρατηρήσή μου αφορά την... καταρχάς ε, να σας ευχαριστήσω που ε, ήρθατε εδώ μαζί μας και δεύτερον ε, ήθελα να πω για την κοινή, για τον κοινό προγραμματισμό. Κάποιος, ένας συνάδελφος μίλησε για τον εξευρωπαϊσμό της έρευνας. Καλό θα είναι να μπορούμε να κάνουμε έναν κοινό προγραμματισμό. Η εμπειρία όμως μας λέει για το Alzheimer, πράγμα το πρώτο, ήταν το πρώτο project, ε, είναι ότι... Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο γιατί ξεκινάμε από ένα πάρα πολύ καμηλό κατόφλι και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε ε, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Τέλος πάντων, αυτό το οποίο ρωτάω είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να αναπτύξουμε και να εμβαθύνουμε κάπως τον κοινό προγραμματισμό. Ίσως να αυξήσουμε την ποσόστοση από πλευράς της Ευρώπης. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσει αυτό το θέμα. Και δεύτερον είναι η κοινωνική καινοτομία. Ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία για την κοινωνική καινοτομία και θέλω να ξέρω τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιες και πρωτοβουλίες μπορούν να αναλυφθούν, και η κοινωνική καινοτομία μπορεί να είναι χρήσιμη και για την οικονομική ανάπτυξη, για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων και απέναντι στους εργαζόμενους μπορεί να είναι καλύτερη. Επίσης η διαφοροποίηση των κονδυλίων, το γεωργία, ταμείο συνοχής, ερθωτικά ταμεία, όλες αυτές οι χρηματοδοτήσεις, οι πηγές μάλλον χρηματοδότησης, πώς μπορούν να συνεργαστούν, πώς μπορούν να συνδυαστούν έτσι ώστε να έχουμε ένα πλαίσιο αναφοράς, γιατί και τα, ποσά από το Ταμείο την συνοχή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για, για την καινοτομία και την τοπική ανταγωνιστικότητα. Αλλά θα πρέπει να, είμαστε, να συνδυαστούμε, έτσι ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη και να μην υπάρχει διασπάθηση των κοινοτικών κονδυλίων. Ευχαριστώ. Κύριε Στόιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. <clears throat> Το δικό μου ερώτημα αφορά την αξιολόγηση του έκτου προγράμματος πλαισίου επί τη βάση και επίσης την, το, την ενδιάμεση, για την ενδιάμεση έκθεση του εβδόμου ου προγράμματος πλαισίου. Δεν έχετε μετάφραση. Στο έκτο πρόγραμμα πλαίσιο έγινε σαφές ότι πέραν της υποστήριξης των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων 20% των ε, ε, κονδυλίων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν λειτουργήσαν ουσιαστικά, δεν απορροφήθηκαν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τονίσει ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει υποστήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη για τα ερευνητικά θέματα. Επίσης υπήρχε πιο εύκολη πρόσβαση και στα μέσω των διαχρονικών ταμείων εγώ ήμουν ακριβώ εισηγητή για τα θέματα αυτά υποστήριξη τη έρευνα από τα διαδοτικά ταμεία, αλλά θα, το ερώτημά μου είναι κατά πόσο η Πολυνοϊκή Προεδρία θεωρεί ότι η συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι ένα από τα κέρια σημεία τη πολιτική σα σε σχέση με την έρευνα. Ευχαριστώ. Μπορώ τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Υπουργό. Έχουμε 15 λεπτά μονάχα στη διάθεσή μας και ήταν τόσο πολλές και τόσο δύσκολες ερωτήσεις. Ελπίζω ότι θα προσπαθήσετε να τις απαντήσετε όλες. Um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους για τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. που δείχνουν πόσο διαφορετικές προκλήσεις έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο ερωτήσεις. Είναι πράγματα που με ρώτησαν η κυρία Καρβάλιο και ο κύριος Μαρτσινκέβιτς. Και αυτό γιατί επικαλύπτονται λιγάκι δύο αυτές ερωτήσεις μεταξύ τους. Είναι και δύο ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με την πολιτική απλοποίηση και οι δύο αναφερθήκατε στην αναγκαιότητα να βρούμε νέους τρόπους χρηματοδότησης, νέες ευκαιρίες για χρηματοδότηση. Όταν μιλάμε για απλοποίηση, είναι αλήθεια ότι εκτιμούμε όλους ιδιαίτερα στην έκθεση της κυρίας ε, Καρβάλιο για την απλοποίηση. Οι 71 συστάσεις ήταν κάτι που εκτιμήσαμε όλους ιδιαίτερα. Είναι πολύ σημαντικές. Ξέρουμε βέβαια ότι δεν είναι πάντα εύκολο να τεθούν σε εφαρμογή οι 71 αυτές οι συστάσεις. Όμως, το βασικό εμπόδιο για την αριστεία που είναι η χρηματοδότηση είναι και το πιο δύσκολο πρόβλημα. Αν αυτό μπορούσαμε να το λύσουμε και νομίζω ότι θα το κάναμε αυτό ακριβώς απλοποιώντας. Και εφόσον οι ετούντες ήταν αντιμέτωποι με πιο απλοποιημένες διαδικασίες. Αυτό θα βοηθούσε και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με την Προεδρία μας, να μην υπάρχουν οικονομικά εμπόδια. Καταλήξαμε σε κάποια συμπεράσματα, μεταξύ των οποίων ένα νέο υπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη μας τα καταποκοπή ποσά, έναν υπολογισμό καταποκοπή, οπότε πιο ταλαντούχοι ερευνητέ και επιστήμονες να μπορούν να ξεκινούν το έργο τους. Γιατί έτσι θα μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα επικεντρωθούμε στην άρση των ε, εμποδίων, ό,τι είδους και αν είναι αυτά, Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και μια τάση για αναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι μια εναρμόνιση και των δαπανών και του προγράμματος. Υπάρχει λοιπόν προσπάθεια εναρμόνισης. Και τώρα έρχομαι σε μια άλλη ερώτηση που μου κάνατε. Έχουμε την εντύπωση και ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε ενιαίες διαδικασίες παντού και σε όλα. Αν όμως καταφέρουμε και αναπτύξουμε κάποιους κανόνες που μεταξύ τους να ευθυγραμμίζονται. Κανόνες για παράδειγμα για την αξιολόγηση των προγραμμάτων. Ήδη αυτό θα είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δε ποσά τα οποία προορίζονται για την έρευνα και την καινοτομία θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Η χρηματοδότηση γίνεται από τα διορθωτικά ταμεία και από το πρόγραμμα πλαίσιο επιπλέον έχουμε και πόρους εθνικούς από τα κράτη-μέλη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε οι διαδικασίες αυτές να ευθυγραμμίζονται πολύ περισσότερο μεταξύ τους και οι νέες διαδικασίες, το νέο πρόγραμμα να είναι πιο απλές και πιο εύκολα εφαρμόσιμες. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι τα κράτη-μέλη πάντα έχουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν. Εννοείται ότι υπάρχουν τα μέσα τα οποία από τη φύση τους συνδυάζουν την χρηματοδότηση προγραμμάτων και από τα προγράμματα πλαίσιο και από άλλες οικονομικές πηγές, εθνική πόρη για παράδειγμα. Γι' αυτό και εδώ θέλω να έρθω στην ερώτηση που έκανε η κυρία Τόγια. Η ερώτηση είχε να κάνει με ένα θέμα σχεδιασμού της χρηματοδότησης της έρευνας στην πρωτοβουλία των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί ευρέως Θα συζητηθεί δηλαδή στις συνεδριάσει του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο για παράδειγμα σε ένα επίσημο συμβούλιο που θα γίνει εδώ στις Βρυξέλλες. Εκεί θα συζητηθεί αυτό το θέμα. Και αυτό γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι πρέπει να βρίσκουμε τέτοια μέσα και να χρησιμοποιούμε τέτοια μέσα τα οποία από τη μια μεριά μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε καλύτερα τον κοινό σχεδιασμό και προγραμματισμό και από την άλλη μεριά θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ε, γενικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Τέτοιες πρωτοβουλίες από κάτω προς τα πάνω μπορούν να εφαρμοστούν λαμβάνοντας υπόψη τις παγκόσμιες προκλήσεις. Είμαι σίγουρη ότι τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εμπειρία από τέτοιον κοινό προγραμματισμό. Συγχρόνως τα κράτη-μέλη μπορούν έτσι να χρησιμοποιήσουν και άλλους οικονομικούς πόρους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως προτείνει κάποιες ιδέες για παράδειγμα, έχει εντοπίσει κάποιες παγκόσμιες προκλήσεις και για το Συμβούλιο η αξιολόγηση της πρώτης πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης για την ε, υγιή γύρανση θα αποτελέσει μια κατευθυντήρια γραμμή για το τι να κάνουμε στη συνέχεια, για το κατά πόσο δηλαδή πρέπει να αναπτύξουμε τα προγράμματα που έχουν ε, εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του μέσου για την εταιρική σχέση για την καινοτομία. Πρόκειται για θέματα, για παράδειγμα, αγροτικής πολιτικής. Στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, χωρίς τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του πρώτου προγράμματος που έχει να κάνει, όπως είπαμε, με ε, την υγιή γύρενση. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του Συμβουλίου. Πάντως, η Πολωνική Προεδρία θα προσπαθήσει να πετύχει συνένεση. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να προχωρήσουμε στις καλύτερες δυνατόν διαδικασίες ώστε να έχουμε ένα συντονισμό ε, τη έρευνα μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνού επίπεδου. Υπήρξαν και άλλε ενδιαφέρουσε ερωτήσει που μου κάνατε για την πολιτική καινοτομία, στη σχέση τη καινοτομία με την οικονομία. Ή άλλο παράδειγμα, ο κύριος Γκέρεκ προτείνει να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό πάνελ το οποίο να αναλύει όλες τις θεωρίες που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Θα μπορούσαμε όντω, μέσω κοινού προγραμματισμού ή μέσω άλλων δραστηριοτήτων να δουλέψουμε πάνω σε διαφορετικές ενεργειακές πολιτικές μέσω εταιρικής σχέσης για την καινοτομία. Συνεπώς, πιστεύω ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας ότι πολλά ερευνητικά αποτελέσματα καθόλου παρά άριστα είναι. Και τέτοια αποτελέσματα μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα όταν προχωράμε στην εκπόνηση πολιτικής. Κύριος στόχος λοιπόν είναι να έχουμε μια εναρμονισμένη οικονομική ανάπτυξη ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Για τον κύριο Μάρση τώρα. Με ρωτήσατε κι εσείς κάτι. Νομίζω ότι ήδη αναφέρθηκα στην απλοποίηση και αναφέρθηκα στη συνέργεια με το Ταμείο Συνοχής. Όπως επίσης και με οριζόντια προγράμματα. Πάντως είναι ζωτική σημασίας να προσθέσω το εξή Για μας Οι υποδομές για την έρευνα και η ανάπτυξή τους είναι πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την πρώτη διπουργική διάσκεψη και μετά θα ακολουθήσει η συνεδρία του Συμβουλίου. Κατά τη διάσκεψη αυτή λοιπόν θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις μεγαλύτερες αδυναμίες. Θα προσπαθήσουμε επίσης να εντοπίσουμε και τα δυνατά σημεία του συστήματος ώστε ώστε να έχουμε υπόψη μας και την περιφερειακή διάσταση. Θέλουμε να έχουμε μία πολιτική ανάπτυξης, μία ευφύ πολιτική που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορές των διάφορων περιφερειών, τα δύνατα και τα δυνατά του σημεία, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται και τις υποδομές που έχουν στη διάθεσή τους ή που πρέπει να δημιουργηθούν στον κοις μέλλον. Τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να τις συντονίζουμε τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο. Μόνο έτσι δεν θα επαναλαμβάνουμε τις ίδιες δραστηριότητες χωρίς λόγο, δεν θα υπάρχει επικάλυψη επίσης υποδομών. Ένα άλλο θέμα είναι να επιτρέψουμε στους νέους επιστήμονες να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και αυτοί οι νέοι επιστήμονες να είναι από όλες τις χώρες μέλη. Ξέρω ότι πρέπει να τελειώσω. Αλλά συμπληρώνω το εξής. Έχουμε εμπειρίες από το παρελθόν για υποδομές που πρέπει να είναι στη διάθεση των νέων. Κύριε Γιόγκρισαν επίσης ρώτησε κάτι για το πώς θα αξιολογήσουμε το ερευνητικό δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας και τι θα κάνουμε με την ανεργία των νέων στην Ευρώπη. Υπάρχουν διαφορετικές μετρήσεις για το ερευνητικό δυναμικό στην Ευρώπη που κάθε άλλο παρά Τέλεις είναι. Ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με ένα νέο κριτήριο προκειμένου να είμαστε σε θέση να υπολογίζουμε το βαθμό καινοτομία. Και σε αυτό το βαθμό καινοτομία πρέπει να μπορούμε να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο για να δούμε πού βρίσκεται η αποτελεσματικότητα στην ε, καινοτομία, η αποτελεσματικότητα των ε, εθνικών ε, και των ευρωπαϊκών πόρων, που είναι η προστιθέμενη αξία δηλαδή των πόρων. Γιατί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι η έρευνά μας να καταλήγει σε καλύτερα προϊόντα και σε καλύτερες υπηρεσίες. Αυτό μας ενδιαφέρει, γι' αυτό τι θέλουμε την έρευνα και την καινοτομία. Άρα είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε για τη βασική έρευνα, τη θεμελιώδη έρευνα, ε, πού βρίσκεται το ερευνητικό δυναμικό στην Ευρώπη. Και τέλος για την ανεργία στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που είχαμε ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θα σας μεταφέρω κάποια προσωπική εμπειρία που έχω από την Πολωνία. Στην Πολωνία χρησιμοποιήσαμε τα διευθυντικά ταμεία για να στηρίξουμε αυτούς που θέλουν να σπουδάσουν, για να στηρίξουμε τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν ακριβείς επιστήμες, τεχνολογία. Γιατί όντως πολλές θέσεις απασχόλησης είναι διαθέσιμες γι' αυτό, γιατί έχουμε στην ανεργία νέους από τα πανεπιστήμια με κάποιες επιστημονικές γνώσεις, αλλά αυτοί που σπουδάζουν για να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές θα έχουν λιγότερη δουλειά στο μέλλον, γιατί όλο και λιγότεροι δάσκαλοι και καθηγητές θα χρειάζονται. Γι' αυτό λοιπόν τώρα τα ιδιωτικά ταμεία τα χρησιμοποιούμε για να οργανώσουμε σπουδές και να στηρίξουμε σπουδές στις ακριβείς επιστήμες που πιστεύουμε ότι θα οδηγήσουν τους φοιτητές σε επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας λοιπόν όταν μιλάμε για έρευνα, να ξέρουμε τι τεχνολογίες θα χρειαστούν, τι γνώσεις θα χρειαστούν, ώστε οι φοιτητέ που θα τελειώσουν τέτοιου είδου σπουδέ να μπορούν να βρουν δουλειά. Πρέπει να αναλύουμε τι ανάγκε τη αγορά εργασία, λοιπόν. Οι επιχειρηματίε πολλέ φορέ λένε ότι να, δεν χρειάζονται περισσότεροι δάσκαλοι, περισσότεροι καθηγητέ, αυτοί που χρειάζονται είναι μηχανικοί ή ειδικοί για την πληροφορική κτλ. Τέλος πρέπει να απαντήσω ακόμα και στην ερώτηση του κύριου Τάιρερ, ο οποίος ρώτησε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ίσως να μην έδωσα αρκετή σημασία στην αρχή, αλλά όντω είναι μια από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες της πολωνικής προεδρίας. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά και ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η συμμετοχή των ε, μικρών ερευνητικών μονάδων, αλλά και η συμμετοχή και των φοιτητών ε, βέβαια αυτών που μόλις παίρνουν το πτυχίο τους αλλά και των ε, μικρών επιχειρήσεων, ε, των start που βρίσκονται στην αρχή. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε έχοντας τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή μας μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε την οικονομία μας και έτσι θα προσελκύσουμε και περισσότερη καινοτομία. Βλέπω τον πρόεδρο αρχίζει να εκνευρίζεται. Έχω μιλήσει υπερβολικά πολύ φαίνεται. Οπότε θα σταματήσω εδώ. Αν δεν κάλυψα όλες σας τις ερωτήσεις, είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και ευχαρίστως να απαντήσω και αργότερα. Δεν απάντησα όμως στην κυρία Κολάσκα Βομπίνσκα για αυτό που είπε. Θα το κάνω πολύ σύντομα. Φυσικά και υπάρχουν πολλές ιδέες για το πώς μπορούμε να λύσουμε το θέμα της ε, λιγότερης εκπροσώπησης, της μικρότερης εκπροσώπησης ορισμένων χωρών ή περιφερειών εξαιτίας των κριτηρίων αριστείας. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει κάποια συμπεράσματα από την αξιολόγηση, από την ανάλυση που θα κάνει όσον αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για την έρευνα. Και βάσει των συμπερισμάτων αυτών θα καταλήξουμε σε νέες ιδέες που έχουν να κάνουν με την ε, ανάλυση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ που με καλέσατε εδώ. Πρέπει να σας ομολογήσω ότι προσωπικά για μένα αυτό με φέρνει σε παλιούς καιρούς πριν από χρόνια που ήμουν βέβαια στα έδρανα και όχι εδώ στο Προεδρείο, τότε που ήμουν Ευρωβουλευτής κι εγώ. Σας ευχαριστώ που μπόρεσα να σας συναντήσω και να σας μιλήσω αυτή τη φορά από το Προεδρείο. Και για μας ήταν μια εξαιρετική εμπειρία κυρία Υπουργέ. Χαρήκαμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Αλλά θα σας ξαναδούμε μέσα σε αυτό το εξάμεινο της πολιτικής ε, προεδρίας. Γι' αυτό σας ζητούμε την κατανόησή σας γιατί έχουμε πίεση χρόνου σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν θαυμάσια πάντως αυτά τα οποία ακούσαμε από εσά. Ευχαριστώ πολύ. 4 okay? Anna, we need some time. Oh, yeah, technique. Sometimes it's complicated. Meine Damen, meine Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen. Κυρίε και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, μπορώ να κάνω κάποιε εισαγωγικέ παρατηρήσει. Καταρχήν, να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργούν τα, τα διερμηνευτικά μηχανήματα. Νομίζω ότι λειτουργούν πλέον. Σήμερα και αύριο έχουμε πολλούς συνομιλητές και πρέπει να κανονίσουμε και την χρονική τους ε, την χρονική ρύθμιση για όλες αυτές τις επαφές. Θα ήθελα να σας πω τώρα ότι ο Διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενεργείας, ο κύριος ε, Τάνα, Τανάκα, ήρθε ενώπιόν μας. Θέλω να τον ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας και, και εξ ονόματος της Επιτροπής μας. Ξέρουμε όλοι ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα να αντιμετωπίσετε, πάρα πολλά προβλήματα να επιλύσετε, αλλά ξέρετε ότι και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια μέσα στα πλαίσια του ενεργειακού μείγματος στην Ευρώπη, την τροφοδοσία της Ευρώπης σε, ενέργεια. Μετά από την πυρηνική λοιπόν καταστροφή στην Φουκουσίμα έχουν υπάρξει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης μας στην Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν όχι μονάχα να ε, υπάρχει ο συγκλονισμός που νιώσαμε όλοι, αλλά να ακούσουμε και τις απόψεις και τις ιδέες που θα μπορούσατε να μας δώσετε. Θα χαρούμε πάρα πολύ να πάρουμε οποιασδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που θα μας βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήλθατε και δεν θα μακρηγορήσω, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να έλθω και πάλι ενώπιον της Επιτροπής σας και να παρουσιάσω την ε, ανάλυση της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας. Όπως τα ξέρετε, η αποστολή του οργανισμού μας, ο οποίος έχει έδρα το Παρίσι, είναι να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της παραγωγής ενέργειας. Και ο βασικός μας ε, στόχος καταρχήν ήταν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, το εξασφαλίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ώστε να εξασφαλίσουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η αγορά λόγω της διαταραχής μετά τα γεγονότα στην αγορά πετρελαίου, μετά τις αλλαγές, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Λιβύη. Φυσικά θα απαντήσω οποιοδήποτε ερώτημα έχετε για τα θέματα αυτά, αλλά σήμερα θα ήθελα να εστιάσω πολύ περισσότερο την ε, παρέμβασή μου στον αντίκτυπο του ατυχήματος της Φουκουσίμα και όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για μια καταστροφή, ένα γεγονός ολέθριο το οποίο έχει τεράστιο αντίκτυπο σε όλο τον τομέα ενέργειας και ιδίως σε σχέση με το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας. Ως ε, Ιάπων και εγώ προσωπικά νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη για το ατύχημα αυτό που το είναι τώρα στο δρόμο της σταθεροποίησης, αλλά θέλω επίσης και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη για τη βοήθεια που δώσαν οι κυβερνήσεις από όλο τον κόσμο για να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες του τσουναμιού και του σεισμού και φυσικά όχι μοναχά της πυρηνικής καταστροφής. Εμείς τώρα βρισκόμαστε στο δρόμο της ανοικοδόμησης και της αποκατάστασης. Πολλές οικονομικές δραστηριότητες επανέρχονται στην Ιαπωνία. <clears throat> Είμαι απόλυτα πεπισμένος και Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα ανακάμψει μετά από αυτή την καταστροφή η Ιαπωνία. Τούτου λεχθέντος. Η, Επιτροπή, η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας έχει προβεί και προβαίνει ακόμα σε μία ανάλυση την λεγόμενη δημιουργία σεναρίων που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό σε σχέση και με τα θέματα στρατηγικών αποθεμάτων. Αν δεν ξέρει κανείς μια αγορά, είναι πολύ δύσκολο να ξέρει πόσο πετρέλαιο χρειαζόμαστε, πόση ενέργεια θα μας λείψει, τι είδους πολιτικές ε, συστάσεις μπορούμε να κάνουμε στα κράτη-μέλη μας ή ακόμα και σε μεγάλους καταναλωτές ενέργειες που δεν ανήκουν στην ε, Διεθνή Επιτροπή, ε, στο Διεθνή Φορέα Ατομικής Ενέργειας. Το 2011 λοιπόν θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο θα είναι από τα σημαντικότερα θέματα που θα αντιμετωπίσουμε. Αυτά τα οποία θέλω να σας πω σήμερα είναι ένα είδος πρόγευσης αυτού που θα συζητήθει για τα πυρηνικά θέματα. Να σας παρουσιάσω τώρα ποια είναι η τωρινή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος είναι ο πραγματικός λόγος για την καταστροφή στη Φουκουσίμα. Θα χρειαστεί να αναμείνουμε να υπάρξει η πλήρης ανάλυση που θα γίνει από τις Ιαπωνικές Αρχές και τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας για το τι πήγε στραβά. <clears throat> να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με πρόληψη κινδύνου, τα προβλήματα αρχιτεκτονικής των πυρηνικών σταθμών, Όλα αυτά λοιπόν είναι ζητήματα τα οποία δεν θα έχουν διαλευκανθεί οριστικά παρά μόνο όταν έχουμε την οριστική έκθεση. Αλλά πιστεύω ότι μετά από τη σταθεροποίηση του τον πυρηνικό σταθμό στη, στη Φουκουσίμα, θα έχουμε αποκομίσει τα απαραίτητα διδάγματα και θα έχουμε ενισχύσει τις γνώσεις μας σε σχέση με την πυρηνική τεχνολογία. Είδαμε λοιπόν το σημαντικό ρόλο που είχε η πυρηνική ενέργεια στο ενεργειακό μείγμα του μέλλοντος. Μετά όμως το ατύχημα της Φουκουσίμα είναι γνωστό ότι κάποιες χώρες στην Ευρώπη αλλά και αλλού άρχισαν να αναθεωρούν τη θέση τους σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Οι προηγούμενες λοιπόν προβλέψεις, τα προηγούμενα σενάρια της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ξαφνικά αυτή τη στιγμή φαίνονται υπερβολικά ρόδινα και αισιόδοξα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας και τα σενάριά μας και να προσαρμοστούμε στην, ε, στον απόϊχο της ε, Φουκουσίμα. Φυσικά η ανάπτυξη νέων μορφών ενέργειας θα γίνει με βαδί ε, ρυθμό και φυσικά ξέρουμε ότι στο άμεσο και απότερο μέλλον θα κλείσουν και πολλοί πυρηνικοί σταθμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλού. Αναλύουμε λοιπόν την κατάσταση και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και υπάρχουν ε, σε χώρες όπως είναι η Ελβετία, η Ιταλία, φυσικά η Γερμανία, πολλές ανησυχίες αυτό είναι σαφές, αλλά είναι επίσης σαφές ότι, όπως δίνει και η επόμενη διαφάνεια, υπάρχει σημαντική δέσμευση ακόμα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης όπως φυσικά η Ρωσία, η Νότια Αφρική, η Ινδία και η Κίνα που εξακολουθούν να είναι προσιλωμένε στη χρήση τη πυρηνική ενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν ανάμεικτε απόψεις σε σχέση με την πυρηνική ενέργεια. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να έχουμε κάποιες υποθέσεις επί των οποίων να εδράσονται τα σενάρια μας. Και η, το σενάριο με το οποίο λειτουργούμε είναι ότι τα υποκατασκευή πυρηνική σταθμή θα αυτοί που είναι υποκατασκευή θα περατωθούν, ενώ στις χώρες του ΟΣΑ τουλάχιστον θα υπάρξει πολύ βραδύτερη ανάπτυξη νέων πυρηνικών σταθμών. Και φυσικά εμείς επί τη βάση αυτού του σενάριου υπολογίζουμε τι σημαίνει αυτό σε σχέση με τις συνολικές τάσεις για την παγκόσμια παραγωγή πυρηνική ενέργεια, τι σημαίνει για το τίμημα τη κιλοβατόρα, τι σημαίνει σε επίπεδο παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, σε σχέση με το παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα, πώ θα μπορέσουμε επίση να αντιμετωπίσουμε και την κλιματική αλλαγή και τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, συγκεκριμένα διοξιδίου του άνθρακο. Επομένω λοιπόν όλα αυτά τα σενάρια <clears throat> και φέτο και του χρόνου θα οδηγήσουν σε μια πιο ενδελεχή αντιμετώπιση κατά χώρα, μια πιο προσεκτική ανάλυση για τα νέα αυτά σενάρια που βασίζονται σε χαμηλότερη χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα, για τις υποθέσεις τις οποίες έχουμε σαν υποθέσεις εργασίας. Αν οι αναπτυγμένες οικονομίες του ΩΣΑ μειώσουν την ε, ανάπτυξη της ε, πυρηνικής ενέργειας, ενώ οι χώρες που δεν είναι στον ΩΣΑ διατηρήσουν κάποιους από τους πυρηνικούς σταθμούς τους τουλάχιστον, αν όχι περισσότερους, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα προσθήκης νέων μονάδων στο ποινικό τομέα θα είναι το μισό από αυτά που περιμέναμε στο λεγόμενο σενάριο νέων πολιτικών. Ήταν ένα σενάριο αυτό το οποίο προέβλεπε κάποιες αυξήσεις σε πυρηνική δυναμικότητα, παίρνει την ε, πιο, τη λιγότερο φιλόδοξη πλευρά των συμφωνιών της Κοπερχάγης είναι πιο δύσκολο να πετύχουμε το σενάριο των δύο βαθμών μονάχα αύξηση θερμοκρασία, δηλαδή το σενάριο των 450 μερών ανά εκατομμύριο για το διοξίδιο του άνθρακο, αλλά το σενάριο αυτό χαμηλών φιλοδεξιών περιμένουμε ότι 360 γίγαβατ πρόσθετης παραγωγικής ικανότητος θα είναι απαραίτητα και θα κατασκευαστούν. Αυτό φυσικά περιλαμβάνει και την αντεκατάσταση των γυρασκών των πυρηνικών σταθμών. Και στο σενάυτο σενάριο κατεβαίνουμε από τα 360 πρόσθετα γίγαβατ σε 180 πρόσθετα γίγαβατ, τα οποία υποθέτουμε ότι θα κατασκευαστούν στο χαμηλότερο αυτό πυρηνικό σενάριο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει σχεδόν μια σταθεροποίηση της πυρηνικής ικανότητας, παραγωγικής ικανότητας μέχρι το 2035. Και το, το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας θα κατέβει από 14% που είναι τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο σε 10% ποσοστό της συνολικής παραγωγής ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν σε σχέση με το, με το τίμημα των, με τις τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος. Υπάρχει επίσης και αντίκτυπο σε άλλους τομείς. Εμείς απλώς θεωρήσαμε ότι η ικανότητα που θα χαθεί για την πυρηνική ενέργεια σε ό,τι αφορά την ηλεκτροπαραγωγή θα αντικατασταθεί κατά ένα τρίτο από άνθρακα, ένα τρίτο από φυσικό αέρα, ένα τρίτο από ανανεώσιμες ενέργειες. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικά διαφορικά κόστους, αλλά η πρόβλεψή μας είναι ότι κάθε ένας από αυτούς τους τρεις τομείς θα καλύψει το ένα τρίτο των αναγκών που θα δημιουργηθούν με τη μείωση της ε, πυρηνικής ενέργειας Επομένως αυτό θα οδηγήσει σε εκπομπή 130 εκατομμυρίων ε, ισοδυνάμου άνθρακος. Το 2035 δηλαδή ουσιαστικά θα πρέπει να έχουμε μία ακόμα Αυστραλία σε ό,τι αφορά ηλεκτρισμό από άνθρακα. Δύο δισεκατομμύρια λίτρα παραγωγή φυσικού αερίου θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε ένα πρόσθετο κατά λοιπόν σε παραγωγή φυσικού αερίου μέχρι το 2035. Για τις ανανεώσιμες ενέργειες 460 εκατομμύρια κιλοβατόρες μέχρι το 2035, πέντε φορές δηλαδή, την ε, ανανεώσιμη ενέργεια που παράγεται στη Γερμανία σήμερα. Πέντε ανανεώσιμες Γερμανίες θέλουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν είναι ο αντίκτυπος του σενάριου που σας ανέφερα, το χαμηλό πυρηνικό σενάριο και αυτές είναι οι πρόσθετες ανάγκες για παραγωγή από άνθρακα, φυσικό αέριο και ανανεώσιμες ενέργειες. Όλα αυτά αναπόφευκτα σημαίνουν υψηλότερε τιμές άνθρακος, φυσικού αερίου και ανανεωσίμων ενεργειών. Φυσικά αν υπάρξει μαζική ανάπτυξη θα μειωθεί το κόστος, αλλά οι ανανεώσιμες ενέργειες είναι ακόμα πολύ δάπανες. Αυτό σημαίνει το κόστος ηλεκτρισμού και τα τέλη ηλεκτρισμού θα ανέλθουν. Η επόμενη διαφάνεια δείχνει ποιες είναι οι προβλέψεις μας για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος. Το... Η στήλη με το ελαφρό γαλάζιο δείχνει τα νέα σενάρια πολιτικής. Ναι, εδώ προβλέπεται να γίνει μια σταθεροποίηση, αλλά όχι να υπάρξει μείωση στο βαθμό που θέλουμε να πετύχουμε για να διατηρηθεί το σενάριο των δύο βαθμών αύξησης θερμοκρασίας μονάχα. Σε σχέση με αυτό το νέο σενάριο πολιτικής, λόγω της χρήσης φυσικού αερίου και άνθρακος, αυτό το νέο σενάριο 0,5 γιγατόνους περισσότερο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, περίπου 30% περισσότερο εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος από τον τομέα παραγωγής ισχύω το 2035, που θα πρέπει να προσθεθούν στην αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος μεταξύ 2010-2035. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, αυτό μειώνει κατά δύο αυτά τα οποία, κατά, στο ένα δεύτερο αυτό το στόχο της, του μετριασμού που θέλαμε να πετύχουμε. Δηλαδή γίνεται πολύ πιο δύσκολος ο στόχος του μετριασμού ως το 2050. Για το 2035 επίσης η ανάπτυξη της διαδικασίας συγκράτησης και αποθήκευσης ε, άνθρακος θα γίνει πολύ σημαντική γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το 2050 για να έχουμε 50% μείωση στην εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος θα χρειαστούμε 50% της ενέργειας να είναι ανανεώσιμες και το άλλο 50% να είναι πυρηνική ενέργεια ή να περιέχει τεχνολογία συγκράτησης και αποθήκευσης του άνθρακος. Λοιπόν, αν μειωθεί τόσο έντονα η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να επενδύσουμε μαζικά στη συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακος και αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο για τον καθορισμό των τιμών άνθρακος. Αυτά λοιπόν παρουσιάζει η ανάλυση μας για τη Γερμανία. Γιατί η Γερμανία έχει πάρει μια φιλόδοξη απόφαση μέχρι το 2022 να κλείσει όλους τους ποινικούς σταθμούς της. Και αν πραγματοποιηθεί αυτή η πολιτική, αυτό θα σημαίνει, θα σημαίνει και αν η Γερμανία μειώσει κατά 10% την κατανάλωση ενέργειας, δηλαδή να αυξήσει την αποδοτικότητα ενέργεια, ενώ συγχρόνως διατηρεί την ε, ε, ένταση ενέργειας και αυξάνει συγχρόνως την ε, οικονομική της ανάπτυξη, τότε το μαύρο τμήμα του γραφήματος θα εξαφανιστεί και θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα φιλόδοξο στόχο 35% ανανεώσιμες ενέργειες και αυτό σημαίνει ότι η Γερμανία θα πρέπει να μειώσει σημαντικά τη χρήση άνθρακος για να κρατήσει τους στόχους θεωρία θερμοκηπίου ενώ θα πρέπει να αυξήσει άλλες μορφές παραγωγής ενέργειας με φυσικό ε, αέριο και αυτό θα σημαίνει δισεκατομμύρια ε, κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ως εισαγωγή αυτό ευχαριστεί μεν την Ρωσία, αλλά δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα ασφάλεια εφοδιασμού, όχι μόνο για τη Γερμανία, αλλά για όλη την Ευρώπη, γιατί γνωρίζουμε ότι το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού έχει πολύ καλή διασύνδεση και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σύνολο με τη χρήση μεγαλύτερης, μεγαλύτερου ποσοστού ανανεώσιμης ενέργειας μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού και το έντονα διασυνδεδεμένο δίκτυο είναι μία από τις βέλτιστες πρακτικές σε όλο τον κόσμο. Αλλά βλέπετε ότι μία απόφαση μιας χώρας και μοναχά, μια σημαντικής χώρας όπως η Γερμανία, μέσω του διασυνδεδεμένου αυτού δικτύου θα έχει σημαντικό αντίκτυπο και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένω, ναι, λέμε, η Γερμανία είναι μία χώρα η οποία είναι κυρίαρχη, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η απόφαση της ως κυρίαρχης χώρας, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να υπάρξει πολύ καλή μορφή συντονισμού μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί υπάρχει αντίκτυπος και στα άλλα κράτη-μέλη. στο επόμενο, στην επόμενη διαφάνεια. Πού θα κατασκευαστούν οι νέοι πυρηνικοί σταθμοί στο νέο σενάριο πολιτικής. Το νέο σενάριο δεν είναι ένα σενάριο μονάχα χαμηλής πυρηνικής ενέργειας, είναι γενικά ένα νέο σενάριο. Από τώρα στο 2020 το μεγαλύτερο μέρος των σταθμών που είναι υποκατασκευή και υποσχεδίαση αφορά την Κίνα και άλλες χώρες που δεν είναι μέσα στα πλαίσια του ΩΣΑ. Μετά το 2020 θα υπάρξει αύξηση στο γαλάζιο, ε, στη γαλάζια στήλη, στήλη του γραφήματος γιατί θα πρέπει να υπάρξει και αντικατάσταση των ποινικών σταθμών στις χώρες του ΩΣΑ. Το να διατηρήσουμε λοιπόν το επίπεδο αυτό στον ΩΣΑ σημαίνει μεγάλες επενδύσεις οι οποίες θα έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Αλλά στο σενάριό μας χαμηλής χρήσης πυρηνικής ενέργειας μπορεί να μειωθεί στο μισό αυτό το τμήμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη μετατόπιση. Θα υπάρξουν πολύ περισσότεροι πυρηνικοί σταθμοί σε χώρες που δεν είναι χώρες του ΩΣΑ και αυτό σημαίνει και ένα σημαντικό στοιχείο. Υπάρχουν προβλήματα πυρηνική ασφάλειας, προβλήματα πυρην... διάδοσης πυρηνικών όπλων, όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι μόνο σε χώρε του ΟΣΑ, αλλά και σε χώρε εκτό του ΟΣΑ. Αλλιώ η εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης πυρηνική ενέργειας δεν μπορεί να τύχει εγγύησον. Τέλο, κύριε Πρόεδρε, εδώ έχετε ένα γράφημα το οποίο χρησιμοποιούμε για να καταδείξουμε ποιες είναι οι προκλήσεις της βιωσιμότητας. Το σενάριο 450 μερών ανά εκατομμύριο είναι το κάτω μέρος και η κόκκινη γραμμή είναι το λεγόμενο σενάριο business as usual. Τα πράγματα συνεχίζουν όπως έχουν. Η χαμηλότερη γραμμή ήταν το σενάριο για 450 μέρη ανά εκατομμύριο σε διοξείδιο του άνθρακος. Αυτό σημαίνει αύξηση 2 βαθμών Κελσίου μέχρι το 2050. Η μπλε γραμμή τώρα είναι το λεγόμενο σενάριο νέων πολιτικών. Η κόκκινη κουκίδα δείχνει αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι το νέο σενάριο με αύξηση διοξιδίου του άνθρακος λίγο περισσότερο από το σενάριο νέας πολιτικής και έχουμε ένα ακόμα σενάριο το οποίο αναφέρεται χρυσή εποχή του φυσικού αέριου. Το οποίο σημαίνει ότι με την σημαντική αύξηση φυσικού αερίου από τους λεγόμενους ασφαλτικούς χιστόλιθος και με τη μεγάλη ε, ζήτηση που θα υπάρξει στην ε, Κίνα θα υπάρξει πολύ ευρύτερη χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου από ό,τι πιστεύουμε στο προϊόν, στο παρελθόν. Αν πραγματοποιηθεί αυτό λοιπόν το σενάριο υψηλής χρήσης φυσικού αερίου, φυσικά αυτό θα οδηγήσει και πάλι δυστυχώς σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, κάπως λιγότερο από το σενάριο των νέων πολιτικών, αλλά όλα αυτά απέχουν πόρο από τα 450 μέρη ανά εκατομμύριο για το διοξείδιο του άνθρακος. Για να πετύχουμε τα 450 λοιπόν μέρη χρειαζόμαστε ανάπτυξη σε βιοκαύσιμα, σε αποδοτικότητα ενέργειας, σε συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακος. Δεν είναι ανέφικτο αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και εμείς βάζουμε ένα ερωτηματικό, είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθεί το σενάριο των 450 μερών ανά εκατομμύριο. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, αλλά όπως είπα προηγουμένως η ανάλυση μας καταδεικνύει ότι ναι, όταν σκεφτόμαστε για την ασφάλεια της, ε, του βαδισμού σε ενέργεια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις πηγές ενέργειας από κοινού. Δεν μπορούμε αλλιώς να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια της ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια είναι ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγής ενέργειας και εδώ και εμπλέκονται και προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των τροφίμων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν την αποδοτικότητα, την συγκράτηση και αποθήκευση άνθρακος, το φυσικό αέριο, όλα αυτά τα στοιχεία γιατί αλλιώς η ασφάλεια μαζί με τη βιώση, ομότητα στο μέλλον μιας εξισορροπημένης ε, τροφοδοσίας ενέργεια δεν μπορεί να εξασφαλιστεί. Ένα άλλο σημαντικό μήνυμα το οποίο θα σας δώσω είναι ότι η ασφάλεια της ε, ενέργειας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με το πρίσμα το οπτικό μιας χώρας αλλά σε επίπεδο περιφερειακό και το ευρωπαϊκό μοντέλο είναι ένα από τα καλύτερα και γι' αυτό ελπίζουμε ότι η Ευρώπη θα μπορέσει με τις συζητήσεις σας, με τον καθορισμό πολιτική σας και της λήψης αποφάσεων να δείξει το δρόμο και να καταδείξει ότι το μέλλον στην ασφάλεια για την ενέργεια μπορεί να εξασφαλιστεί μονάχα με την καλή διαδικτύωση του δικτύου ηλεκτρισμού στην Ευρώπη, μαζί με ένα πολύ ισορροπημένο τρόπο χρησιμοποίησης των διαφόρων πηγών ενέργειας και συγχρόνως με το να υπάρχει μια ενιαία πολιτική στην Ευρώπη και αυτό ίσως είναι και το κύριο μήνυμα το οποίο θα θέλαμε εμείς να δώσουμε στην Ευρώπη μετά από τη Φουκουσίμα. Ευχαριστώ τα μάλα κύριε Πρόεδρε. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Τανάκα για την ανάλυση σας. Νομίζω πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να συλλέξουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Κυρία Καρβάλη, έχει το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και κύριε Νακάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο σαφή σας παρουσίαση. Μία ερώτηση έχω να κάνω όσον αφορά τον τεχνολογικό οδικό χάρτη βάσει του σεναρίου. Αναφερθήκατε στις διάφορες τεχνολογίες και το CCS πρέπει να είναι όριμο το 2050 με 50% των αντιδραστήρων που θα έχουν αυτή την τεχνολογία τότε. Οι άλλες τεχνολογίες, ποια θα είναι η εξέλιξή τους διότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές ε, αλλαγές χωρίς πυρηνική ενέργεια, τότε η τεχνολογία πρέπει να εξελιχθεί. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους δύο αυτούς στόχους. Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε αυτό παρακαλώ. Κύριε Τανάκα, θέλετε να απαντήσετε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εμείς πιστεύουμε ότι το CCS είναι μία περίπτωση. Εννοείται ότι θέλουμε να δούμε και άλλα πειραματικά, και άλλες πειραματικές μονάδες. Υπάρχει, χρησιμοποιείται και μπορεί να αποθηκευθεί εκεί το υλικό. Μπορεί βέβαια να υπάρξει βελτίωση. αν δούμε και την ε, τιμή του άνθρακα με 50-70, αυτό είναι ένας τομέας πάντως στον οποίο πρέπει να κάνουμε πολλές προσπάθειες. Αλλά όπως λέτε και εσείς υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που χρειάζονται, που είναι αναγκαίες για να υπάρξει αυτή η τεχνολογική επανάσταση. Η ολική ενέργεια χρησιμοποιείται ήδη σε έναν βαθμό. Χρειάζονται και ηλιακή ενέργεια όμως με τα φολτοβαϊκά Χρειάζονται παρετέρω εξελίξεις στις τεχνολογίες αυτές και χρειάζονται και άλλου είδους τεχνολογίες. Η γεωθερμική είναι κάτι εφικτό, αλλά ακόμα δεν εφαρμόζεται αρκετά. Χρειάζονται καινοτόμε μέθοδοι. Πιστεύουμε επίσης ότι είναι σημαντικό να είναι τεχνολογία από την πλευρά του χρήστη ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και από τις μεταφορές, δηλαδή μεταφορές να γίνονται με ηλεκτρικά οχήματα για παράδειγμα. Και τέτοιου είδους τεχνολογία χρειάζεται για να μειωθούν οι εκπομπές. Χρειαζόμαστε επίσης την τεχνολογία του Smart Grid για να αντιμετωπίσουμε την αστάθεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην αγορά εναλλακτικών πηγών ενέργειας έτσι ώστε να έχουμε μια μεγάλη αγορά ε, με διασυνδέσεις. Η διαχείριση μιας τέτοιας αγοράς είναι κάτι πολύ σημαντικό, γι' αυτό και χρειάζεται η τεχνολογία ε, των πληροφοριών. Επιπλέον υπάρχει για το θέμα της αποθήκευσης. Το hydropooling είναι ένας τρόπος, αλλά οι τεχνολογίες πάντως που μπορούν και αποθηκεύουν την ενέργεια, μπορείτε να αναφέρετε πολλές τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και θα έπρεπε να συνδυαστούν αυτές μεταξύ τους. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε ευελιξία και ελευθερία χειρισμών μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάση. Έχει Ίσως δύο ή τρεις ομιλητές μαζί, ναι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τελευταία παρατήρηση του κυρίου Τάνακα ήταν ότι το σενάριο το 350 ppm είναι αδύνατο. Θέλω να ξέρω την άποψή σας για το τι μπορεί να γίνει ώστε να είναι εφικτό και όχι αδύνατο. Ευχαριστώ. Πολύ καλή ερώτηση λέει ο κύριος Είναι πρακτικά αδύνατο. Υπάρχει ένα ερωτηματικό, διότι από τεχνική πλευράς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως θα πρέπει να δώσουμε πολλά χρήματα και να κάνουμε πολλές επενδύσεις για να συμβεί κάτι τέτοιο. Επίσης πιστεύουμε ότι οι διαπραγματευτές για τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο. Τι εννοούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζομαστε μία προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω και όχι το αντίστροφο. Να ορίσουμε τους στόχους και να κατανείμουμε τους στόχους σε όλα τα κράτη-μέλη. Αλλά λόγω της κατάσταση στην Κίνα, της ε, πολιτικής Ηνωμένες Πολιτείες, ε, αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, τουλάχιστον επί του παρόντος, δεν φαίνεται να λειτουργεί. Εφόσον ισχύει αυτό το οποίο προτείνουμε, είναι, είπαμε, από κάτω προς τα πάνω. Γιατί? Διότι όλες αυτές οι τεχνολογίες, εάν εφόσον κλειδώσουμε τις τεχνολογίες αυτές για τα επόμενα 30-40 χρόνια, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κόστος εκπομπής του διοξιδίου του άνθρακα εάν δεν υιοθετήσουμε και κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Π.χ. ας πούμε, να είμαστε έτοιμοι για αυτά τα ε, ιδέες εγκαταστάσεις συγκέντρωσης, συλλογή και αποθήκευσης ε, ε, διοξιδίου του άνθρακα. Θα πρέπει αυτή η τεχνολογία δηλαδή να ε, την εκμεταλλευτούμε εμπορικά. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε σοβαρά προβλήματα για την επίτευξη των στόχων αυτών μέχρι το 2050. Κάτι άλλο το οποίο τώρα θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι αυτή η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας. Η Κίνα θέλει να χρησιμοποιήσει περισσότερο αέριο, το εννοεί αυτό, διότι ξέρουν ότι το πετρέλαιο δεν θα λειτουργεί για πάντα. Ο άνθρακας είναι βρώμικος, άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουν περισσότερο αέριο έτσι ώστε να έχουν φιλικά προς ε, φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια, αλλά να έχουν και ε, την απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται. Οι Κινέζοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πετρέλαιο και τον άνθρακα όπως κανονικά, και το ίδιο δεν μπορούμε για το φυσικό αέριο, διότι εάν οι Κινέζοι συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλο ένα και περισσότερο αέριο, θα ε, αυξηθεί το κόστος της ενέργειας. Και για να το αντιμετωπίσουν αυτό θα πρέπει οι Κινέζοι να υιοθετήσουν πολλά εσωτερικά μέτρα. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την ε, αλλαγή του κλίματος. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να εξασφαλίσουμε μια βιωσιμότητα. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε κάποιες γνώσεις, να, προχωρήσουμε αυτές τις ε, γνώσεις, τουλάχιστον από του παρόντος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τανάκα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε, λέει ο κύριο Κορέα Ντεκάμπο. Μα ε, βοηθάει πάρα πολύ να σκεφτούμε καλύτερα. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία ερώτηση έχει να κάνει με το τελευταίο γράφημα το οποίο παρουσιάσατε, όπου καταγράφεται έχετε χωριστά την περίοδο μέχρι το 2020 και μετά την περίοδο από το 2020 και επέκεινα μέχρι το 2020 βλέπετε να υπάρχει μια αύξηση της χρησιμοποίησης από την Κίνα της πυρηνικής ενέργειας στον πυρηνικό σταθμό μετά το 2020 φαίνεται να μειώνεται αυτή η χρήση. Νομίζω ότι η εξήγηση που δώσατε ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αλλά σε σχέση με τις χώρες που δεν ανήκουν στον ΩΣΑ, εδώ έχω κάποια μεγαλύτερη αμφιβολία, γιατί μετά το 2020 το γράφημά σας δείχνει μια σημαντική αύξηση της πυρηνικής ενέργειας στις χώρες που είναι εκτός του ΩΣΑ. Αν ακολουθήσω λοιπόν την επιχειρηματολογία σας για την τελευταία απάντηση που θα δώσετε, οι χώρες αυτές που δεν είναι στον ΩΣΑ δεν μπορούν και αυτές να έρθουν να σκεφτούν όπως και η Κίνα και να μετριάσουν την κατανάλωση ε, ενεργειακών πόρων να βρούνε άλλες λύσεις, γιατί η πρόβλεψή σας έχει ένα καταστροφικό χαρακτήρα. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν αν υπάρχει και ένα περιθώριο για άλλες εναλλακτικές λύσεις. Το δεύτερο ερώτημα μου τώρα έχει να κάνει με το παράπονο που κάνατε κατά κάποιο τρόπο για την Ευρώπη η οποία δεν έκανε πιο εγκαίρο την αντικατάσταση στον πυρηνικό σταθμό. Καταλαβαίνουμε όλοι αυτό το θέμα. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχασαν απόλυτα την ε, τεχνογνωσία τους σε σχέση με τα πυρηνικά θέματα, σταμάτησαν να εκπαιδεύουν πυρηνικούς μηχανικούς. Η Ευρώπη κλείστηκε σε μία πραξιδηλίας που ήταν η υποχώρηση στην επικουρικότητα. Μα ξέρουμε ότι κάθε ενεργειακή πηγή μπορεί να περάσει και σε άλλες χώρες. Η Ευρώπη δεν μπορεί λοιπόν να λύσει το πρόβλημα αυτό μονάχα ως επικουρικότητα. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να ρωτήσω από εσάς είναι μπορούμε να ανακτήσουμε αυτή τη τεχνολογική στέρηση. Μπορεί η Ευρώπη να ανακτήσει αυτή την απόσταση που έχει σε ένα πολιτικό πλαίσιο στο τωρινό πολιτικό πλαίσιο. Το επιτρέπει το τωρινό πολιτικό πλαίσιο να ανακτήσουμε το χαμένο χρόνο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το οποίο ρωτήσατε. Αυτό το οποίο έδειξα στο τελευταίο γράφημα, το πρώτο τελευταίο γράφημα συγκεκριμένα, είναι ότι πρόκειται για πρόσθετη παραγωγική ικανότητα. Η θα εξακολουθήσει να αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα, αλλά θα μειωθεί η ταχύτητα αύξησης της προστίκης παραγωγική ικανότητα. Ξέρουμε ότι σιγά σιγά σταδιακά μειώνεται η οικονομική ανάπτυξη τη Κίνα, επομένω η ανάγκη να δημιουργηθούν νέοι σταθμοί ισχύω, μεταξύ των οποίων και πυρηνική, θα μειωθεί στα σταθερά και βαθμία μετά το 2020 και προς το 2035. Λόγω αυτού του σενάριου φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μείωση της πυρηνικής ε, ικανότητος στην Κίνα, αλλά φυσικά η συνολική παραγωγική ικανότητα με πυρηνική ενέργεια θα αυξάνεται στην Κίνα. Σε σχέση τώρα με τις χώρες του ΟΣΑ, αυτό το γράφημα δείχνει ότι θα πρέπει να αυξηθεί και η παραγωγική ικανότητα στις χώρες του ΟΣΑ, όπου υπάρχει ακόμα μία ανάγκη αντικατάστασης. Νομίζουμε λοιπόν ότι ακόμα και για να διατηρήσουμε το λεγόμενο ε, σενάριο της νέας, των νέων πολιτικών ο ΩΣΑ θα πρέπει να επενδύσει μαζικά σε νέα παραγωγική ικανότητα, αλλιώ δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα, την ε, ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό δείχνει αυτό το, σχήμα. Στην χαμηλή χρήση πυρηνικής ενέργειας, το μπλε αυτό γράφημα που λέτε, θα είναι πολύ πιο χαμηλό το επίπεδο αυτό. Εδώ θεωρούμε ότι στο, στο σενάριο της χαμηλής πυρηνικής ενέργειας η ανάπτυξη του ΩΣΑ θα μειωθεί σημαντικά. Για το δεύτερο ερώτημα τώρα. Το θέμα της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας. Ναι, ναι η πυρηνική ενέργεια έχει εδρεωθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά... Αλλά λόγω της παράτασης της ζωής των πυρηνικών σταθμών που ήταν το, το, η επιλογή μέχρι τώρα δεν υπήρξε αρκετή καταστροφή, αρκετή διάλυση πυρηνικών σταθμών. Δεν υπήρχε λοιπόν αρκετή γνώση για το πώς θα πρέπει να γίνει αυτή η κατάλυση των πυρηνικών σταθμών. Αυτό είναι μια νέα σημαντική τεχνολογία ανάπτυξη ξαφνικά Έχουμε πιο μεγάλους πυρηνικούς σταθμούς, έχουμε σταθμούς με μεγαλύτερη πυρηνική τεχνολογία, πιο ασφαλείς τεχνολογίες. Με το να φτιάξουμε λοιπόν νέο πυρηνικό σταθμό, αυτό θα αυξήσει την ασφάλεια για την πυρηνική ενέργεια. Αλλά χωρίς επενδύσεις δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρόκειται λοιπόν αυτό μόναχα για τον πυρηνικό τομέα. Αφορά όλες τις τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας χωρίς ε, επενδύσεις χωρίς να επενδύουμε την καλύτερη <clears throat> τεχνολογία, την ε, τρέχουσα καλύτερη τεχνολογία, δεν θα μπορέσει να υπάρξει ανανέωση. Η ανανέωσή μας λοιπόν για την ενέργεια δείχνει ότι ναι, τέτοιου είδους καινοτομίες γίνονται στην ε, Κίνα, γιατί η Κίνα αναπτύχθηκε οικονομικά τόσο γρήγορα και στην αιωλική ενέργεια και στην ηλιακή ενέργεια και στην πυρηνική ενέργεια <clears throat> που ένα μεγάλο μέρος της πρόσθετης παγκόσμια ζήτηση γίνεται στην Κίνα και μετά από το 2020 θα εξακολουθήσει να γίνεται σε κάποιο μικρότερο βαθμό. Σχεδόν ένα κάθε τέσσερα ή πέντε αυτοκίνητα που πουλούνται παγκοσμίω θα είναι στην Κίνα. Η Κίνα λοιπόν θα είναι ο ηγέτης στην τεχνολογική εξέλιξη σε οποιοδήποτε τομέα ο οποίος συνδέεται με την ενέργεια γιατί εκεί θα δημιουργηθεί η πρόσθετη ζήτηση. Οι χώρες του ΟΣΑ και οι χώρες της Ευρώπης έχουν αυτή την πρόκληση. Πώς θα αντιμετωπίσουν, πώς θα ανταγωνιστούν μια, νέα, μια τέτοια χώρα χωρίς νέες επενδύσεις. Λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Φυσικά οι εταιρείε οι οποίες επενδύουν στην Κίνα <clears throat> δοκιμάζουν και νέες τεχνολογίες. Αλλά το να διατηρήσουν στην περιοχή της Ευρώπης την τεχνολογική ικανότητα χωρίς επενδύσεις για νέες τεχνολογίες και νέες μορφές ενέργειας δεν θα είναι πολύ εφικτό. Βλέπουμε πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες είναι προσιλωμένες στην χρήση ανανεώσιμες ενέργειες και αυτό ίσως είναι ο δρόμος. Πολλές ε, ευρωπαϊκές εταιρείες ηλεκτρισμού μιζάρουν στην ε, ανανεώσιμη ενέργεια. Ίσως αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να πετύχουμε μια ε, ριζική αλλαγή, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να είναι ένα τμήμα αυτής της διαδικασίας. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα κομμάτι της αλλαγής. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται πολύ μεγάλη πίεση, υπό μεγάλη πίεση η πυρηνική ενέργεια, το κατανοούμε αυτό και το δεχόμαστε, αλλά συνολικά για να έχουμε βιώσιμη και ασφαλή αγορά ενέργειας στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε όλες τις επιλογές και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε όλες τις επιλογές ενεργειακού χαρακτήρα. Ο κύριος Βιδάλ Κουάδρας. Yes, thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τανάκα για την ε, τόσο πλούσια παρουσίασή σας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και μας υπενθυμίσατε εξάλλου, το ατύχημα της Φουκουσίμα οδήγησε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία, όπως και μη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες, Ελβετία, να προχωρήσουν σε μεγάλες αλλαγές όσον αφορά την ενεργειακή τους πολιτική και τα σχέδιά τους για πυρηνική ενέργεια. Άλλαξαν λοιπόν Αντί να επεκτείνουν ή να χτίσουν νέα πυρηνικά εργοστάσια, αντίθετα σιγά σιγά να εγκαταλείψουν αυτά που ήδη έχουν. Δύο είναι οι ερωτήσεις μου. Πρώτον, από τις δικές σας γνώσεις, τέτοιου είδους αλλαγές στην πολιτική θα λάβουν χώρα και σε άλλες μεγάλες χώρες του κόσμου, στην Κίνα για παράδειγμα την Ινδία ή τις Ηνωμένε Πολιτείες. Ή έχετε την εντύπωση, οι πληροφορίες σας είναι τέτοιες που μπορείτε να μας πείτε πώς θα συνεχίσουν με την πυρηνική ενέργεια όπως και κατά το παρελθόν. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη τώρα. Πέρα από οτιδήποτε πολιτικές απόψεις που δεν είσαστε εδώ για να συζητήσουμε την πολιτική, δεν είσαστε εσείς που θα μας μεταφέρετε την πολιτική, πολιτικές απόψεις, καθαρά τεχνικά μιλώντας. Ορθολογικά για την ασφάλεια εφοδιασμού, μείωση διοξιδίου του άνθρακα, ανάλυση κόστους κέρδους, ε, προβλεπόμενη εξέλιξη των ενεργειακών αναγκών. Καθαρά λοιπόν, βάσει τέτοιων τεχνικών χαρακτηριστικών, πιστεύετε ότι οι θέσεις αυτές είναι ορθές ή όχι. It question Πολύ πολιτική ερώτησή σας και είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς τεχνικά, τεχνολογικά σε αυτήν. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα πως ναι. Όντως είναι σε ένα μεγάλο βαθμό πολιτικό ζήτημα η πυρηνική ενέργεια και είναι απαραίτητη μια πολιτική διάσταση στις διάφορες περιοχές ή χώρες του κόσμου. Είπατε στην αρχή ποιε χώρες θα ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Ναι, στην Ευρώπη η Γερμανία, η Ελβετία, η Ιταλία αποφασίζουν να μην προχωρήσουν με τα πυρηνικά. Η Γαλλία από την άλλη μεριά εξακολουθεί και μένει στην ισχυρή της θέση υπέρ των πυρηνικών. Η Φιλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι υπέρ και από τις ε, χώρες της ε, Ανατολικής Ευρώπης και εκεί πιστεύουν ότι η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ σημαντικό για την ασφαλειά τους. Ρωσία, για παράδειγμα. Υπάρχει λοιπόν μείγμα στην Ευρώπη. Η Κίνα θα συνεχίσει όσο γίνεται περισσότερο, θα συνεχίσει να χτίζει πυρηνικά εργοστάσια γιατί είναι αναγκαίο για αυτούς. Το ίδιο και η Ινδία, η Ρωσία, η Κορέα είναι ένα άλλο παράδειγμα χώρας υπέρ των πυρηνικών. Η Τουρκία επίσης η Νότια Αφρική συνεχίζει να διατηρεί ανοιχτή αυτή την επιλογή των πυρηνικών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι μια περίεργη περίπτωση κατά πάσα πιθανότητα θα τους είναι δύσκολο να χτίσουν νέα πυρηνικά εργοστάσια. Όμως θέλουν να διατηρήσουν την ε, πυρηνική ενέργεια γιατί αυτό είναι αναγκαίο για την ε, οικονομική τους ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν συνολικά ε, πιστεύουμε ότι η κάθε χώρα πρέπει κυρίαρχα να αποφασίσει σχετικά με την πολιτική της για την πυρηνική ενέργεια, τόσο από πολιτικής όσο και τεχνολογίας. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο για κάποια ομάδα χωρών. Και εδώ η Ευρώπη είναι πολύ σοφή που διατηρεί μια διαφοροποίηση στην πολιτική της. Άλλες χώρες είναι υπέρ της πυρηνικής, άλλες όχι. Συνολικά στην Ευρώπη έχετε ανοιχτές όλες τις δυνατότητες. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ ευθύς απόφαση. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρεί κανείς ανοιχτές όλες τις εναλλακτικέ λύσεις. Σίγουρα πολιτικά είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Τεχνολογικά όμως, τι μπορούμε να πούμε. Οι αποφάσεις για τα πυρηνικά είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να επενδύσει μακροπρόθεσμα. Εφόσον υπάρξει αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική, ναι, όχι, ναι, όχι, ανάλογα με το ποια κυβέρνηση είναι στην εξουσία, είναι κάτι που στέλνει ένα πολύ κακό μήνυμα, στραβό μήνυμα. Και αυτό για όλες τις ενέργειες, όχι μόνο για την πυρηνική και για άλλου είδους ενέργειες. Κανένας δεν θα επενδύει αν αλλάζεται γνώμη κάθε τόσο. Άρα το βασικό είναι να υπάρχει μια σταθερή άποψη στις κυβερνήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να προχωρήσουμε σε μια βασική ενεργειακή πολιτική. Η κυρία Κναβίσκα. Ευχαριστώ πολύ ε, εάν ακολουθήσουμε το σενάριο με περισσότερο φυσικό αέριο. Δεν εξαρτώμεθα όλο ένα και περισσότερο από την Ρωσία και επομένως τι πιστεύετε για αυτό το αέριο σχιστόλιθου, γιατί ξεκινάει η συζήτηση και γίνεται πιο καυτή. Και αυτά τα θέματα θα συζητηθούν το φθινόπωρο στο Κοινοβούλιο. Η δεύτερη ερώτηση τώρα είναι η εξής. Ε, είπατε ότι είναι πολύ σωστή, επενέσατε την ε, ευρωπαϊκή πολιτική και αναφερθήκατε και είπατε ότι η απόφαση της Γερμανίας να κλείσει τα πυρηνικά της εργοστάσια θα ε, επηρεάσει την ενεργειακή πολιτική στην Ευρώπη. Επίπως πιστεύετε ότι θα έπρεπε η Γερμανία πριν προχωρήσει σε οτιδήποτε να έχει διευουλευθεί πρώτα με τους υπόλοιπους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαι καγκελάριος, δεν μπορώ να απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση, αλλά νομίζω ότι η Επίτροπος Ότιντζε είπε ε, ότι η γερμανική αυτή απόφαση θα πρέπει να ζητηθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ή άλλως. Καλό θα ήταν να ήταν πριν, αλλά τουλάχιστον εκ των υστέρων καλό θα είναι να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον αντίκτυπο της γερμανικής απόφασης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως στους γείτονες. Και πολλές φορές για τις γερμανικές χώρες αυτή είναι μια ευκαιρία. Ε, ας πούμε μπορείτε να πληρώσετε, να πουλήσετε συγγνώμη ενέργεια σε πολύ καλή τιμή εφόσον η Γερμανία χρειάζεται ενέργεια. Δηλαδή οι χώρες, ε, οι όμορες της Γερμανίας ε, πρέπει να χαίρονται για την απόφαση αυτή αλλά οι καταναλωτές θα πρέπει να πληρώνουν παραπάνω, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί ακριβώς θα γίνεται εξαγωγή της ενέργειας. Επομένως, οι συνέπειες αφορούν όλη την Ευρώπη, άρα πρέπει να το ζητήσει όλη η Ευρώπη, στην Κομισιόν, στο Συμβούλιο, στον ε, στο Κοινοβούλιο. Τώρα, για αυτό το shell gas, αυτό το αέριο από σχιστόλιθο, του σχιστόλιθου μάλλον, ε, δεν το έθιξα. Έχουμε όμως Ε, υπάρχει και ένα άλλο σενάριο. Μπαίνουμε στην ε, εποχή, στη χρυσή εποχή του, του αερίου. Τώρα πρέπει να θέσουμε κάποια ε, ερωτήματα. Είναι ασφαλές το αέριο, όντως έρχεται αυτή η εποχή. Τώρα, αυτό το αέριο του σχιστολίθου δεν είναι διαθέσιμο άμεσα. Καταρχάς, θα πρέπει να να στηριχθούμε πολύ στο συμβατικό φυσικό αέριο, όπως το Κατάρι, αλλά κάποιες άλλες χώρες. θα πρέπει να δούμε καταρχάς την γεωπολιτική κατάσταση του φυσικού αερίου και μετά να προχωρήσουμε. Δηλαδή είναι στρατηγική η απόφαση για να γίνει διαθέσιμο καταρχάς το αέριο αυτό. Το πρόβλημα είναι τώρα είναι ασφαλές, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, περιβαλλοντικά τουλάχιστον. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητήθηκε στι ΗΠΑ, στη Γαλλία, στη Νότια Αφρική. Στις δημοσιεύσεις μας που μπορείτε να, να κατεβάσετε δωρεάν από το site μας, από το site του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, θα δείτε ότι αυτή η τεχνολογία ε, για την ε, για, την, για τον υγρό κατακαιρματισμό είναι διαθέσιμος εδώ και 6 χρόνια στην εξόριξη και χρησιμοποιείται στην εξόριξη πετρελαίου. Δεν είναι καινούριο όμως, αλλά το πρόβλημα είναι η οριζόντια, που, ότι αυτή σε συνδυασμό με την οριζόντια εξόρυξη χρησιμοποιείται για την εξόρυξη αυτού του αέριου. Τώρα, αυτή όμως η τεχνολογία για τον υγρό κατακαιρματισμό δεν είναι αναγκαστικά επικίνδυνη. Στις Ηνωμένε Πολιτείε όμως αυτή η εξόριξη γίνεται πάρα πολύ κοντά στα αστικά κέντρα και δεν είναι πολύ καλές ε, οι συνθήκες εξόριξης. Επομένως τεχνικά μπορεί να γίνει, να προχωρήσουμε. Όμως θα πρέπει να υπάρχει μια, ένας, ε, να υπάρχουν κανονισμοί, ε, να ρυθμιστούν με λεπτομέρειες όλα, τη, όλα τα στάδια της εξόρυξης και αν συμβούν όλα αυτά μπορούμε να προχωρήσουμε. Όμως το κόστος ενδεχόμενα να είναι πιο ακριβό από αυτό που, είναι, που ισχύει τώρα στις πολιτείες. Και επομένως ε, μπορούμε να πούμε ότι το αέριο του σχιστολίθου μπορεί να είναι ο παράγοντας που θα αλλάξει την κατάσταση. Ε, η Πολωνία έχει, η Γαλλία έχει, η Κίνα το έχει, η Αυστραλία το έχει, η Ινδονησία το έχει. Επομένως, εκεί μπορεί να, ότι εκεί μπορεί να αλλάξει η γεωπολιτική κατάσταση του αερίου. Κύριε Σόντι, σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τανάκα για την παρουσία σας. Μεταξύ ημών, δύο ερωτήματα. Διαβάσαμε στα μέσα ενημέρωσης ότι με τις εξελίξεις, ιδίως τα κλεισίματα των πυρηνικών σταθμών στην Ευρώπη, θα μπορέσουμε. Είναι όπως μετά την, ε, <laughs> όπως μετά την ε, μεγάλη ζέστη έχουμε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, μπορούμε να έχουμε πραγματικά ένα τεράστιο πρόβλημα ελλείψη ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο πρόβλημα είναι το θέμα των πυρηνικών σταθμών και της ε, διάλυσής τους. Έχουμε μια τεχνογνωσία στα θέματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση με την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως με τη συνθήκη Ευρατόμ, να αυξήσουμε την ε, έρευνα για την τεχνολογία διάλυσης των πυρηνικών σταθμών. Γιατί μετά από, τα... μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την πυρηνική τεχνολογία, θα πρέπει να διαλύσουμε τους πυρηνικούς σταθμούς που έχουμε. Έχετε κάποια άποψη σε σχέση με τις τεχνολογίες διάλυσης πυρηνικών σταθμών. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ερώτημά σας αφορά το τι θα γίνει εάν η πυρηνική ενέργεια δεν είναι διαθέσιμη όπως περιμέναμε στο παρελθόν. Ξαφνικά επανέρχονται οι άλλοι κίνδυνοι για τη διαταραχή της τροφοδοσίας με ενέργεια στην Ευρώπη και μέσω της διαδικτύωσης μπορεί πολύ εύκολα να επηρεάσει από τη μία περιοχή την άλλη. Αν λοιπόν η πυρηνική ενέργεια είναι λιγότερο διαθέσιμη, θα έχουμε κινδύνους μεγαλύτερους. Η διακοπή τροφοδοσίας από φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας να έχει μεγαλύτερο επίπεδο ε, προβλημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, γίνεται πιο κρίσιμη η τροφοδοσία με φυσικό αέριο αν δεν υπάρχει αρκετή πυρηνική ενέργεια. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτέ όλε τι ε, επιλογέ, όχι πάντα σε μια χώρα, αλλά τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή. Ναι, είναι πρόκληση η διάλυση των πυρηνικών σταθμών. Χρειάζεται χρόνο. <coughs> δεν είμαι ειδικό στην πυρηνική μηχανική, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ήδη η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί για τη διάλυση των πυρηνικών σταθμών και σε ορισμένου πυρηνικού σταθμού έχει εφαρμοστεί αυτή η τεχνολογία. Δεν είναι λοιπόν ένα σημαντικό πρόβλημα το να σταματήσουμε και να διαλύσουμε ένα σταθμό και να υπάρξει ε, καθαρισμός και ανάκτηση του χώρου. Βέβαια το θέμα της ε, ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό για όλους μας Γι' αυτό θα πρέπει να σχεδιάσουμε <clears throat> προσεκτικά και να αναπτύξουμε τέτοιου είδους τεχνολογίες. Αυτό είναι αναφυσβήτητο. Αλλά η τεχνολογία διάλυσης ποινικών σταθμών δεν είναι το βασικό πρόβλημα της χρήσης ποινικής ενέργειας. Αυτό είναι το δικό μου. <clears throat> Αυτή είναι η δική μου άποψη. Η κυρία Σίσλε έχει το λόγο. Γιόρνταν Σίσλε. Ευχαριστώ κύριε Τανάκα. Θα ήθελα να επανέλθω στο ερώτημα που έκανε ο κύριος Κάβρας. Ε, συγγνώμη. Η γερμανική απόφαση ελήφθη με βάση συγκεκριμένα δεδομένα και μετά τη λήψη της απόφασης προχώρησαν σε νιοθέτηση ενός προγράμματος σταδιακής, σταδιακού κλεισίματος των ε, εγκαταστάσεων αυτό, αυτή είναι ένα, αυτό είναι ένα νέο βήμα, αν θέλετε, στον καθορισμό της ενεργειακής πολιτικής. Μέχρι τώρα στηριζόμαστε μόνο σε τεχνικά θέματα. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται ο κόσμος με αυτό το παράδειγμα, αν θέλετε, της ε, Γερμανίας. Πώς βλέπω από ηθικής πλευράς την απόφαση αυτή. Κοιτάξτε, η ηθική είναι ένας τρόπος για να επιλέξει κανείς τον τρόπο της ζωής του. Και ε, ξαφνικά θα έλεγα ότι ότι με βρίσκει σύμφωνο το γεγονός ότι παίρνουμε κάποια φάση με βάση την ηθική. Τούτου λεχθέντο όμως, είναι ηθικό το θέμα του κλεισίματος των εγκαταστάσεων, των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Εγώ έχω ε, κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο αυτή η τεχνολογία θα πρέπει να κρίνεται με ηθικά κριτήρια. Όντως κάθε τεχνολογία υπόκειται σε ηθικά κριτήρια, σε ηθική κρίση, αλλά διαρωτώ με γιατί η πυρηνική ενέργεια ε, έχει πολιτικοποιηθεί τόσο πολύ και ε, προκαλεί τόσες πολλές συζητήσεις ε, και ηθικά διλήμματα σε σχέση με τις άλλες πηγές ενέργειας. Μετά την Φουκουσίμα βέβαια συμφωνώ ότι μπαίνουμε σε ένα νέο τρόπο σκέψης και παραδέχομαι ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αλλά ταυτόχρονα δεν είμαι επιστήμο, δεν είμαι, είμαι, δεν είμαι θετικός επιστήμων, οικονομολόγος είμαι, δεν είμαι μηχανικός, αλλά διαρωτώ με, μήπως θα, πιο, θα πρέπει να είμαστε πιο πολύ ρεαλιστές στις αποφάσεις που παίρνουμε για, τις, για την ενεργειακή πολιτική γιατί όπως είπα και προηγουμένως, σε μια προηγούμενη ερώτηση, η πολιτικοποίηση θα εμποδίσει τις εμπορικές επενδύσεις. Δεν θα επενδύσει κανείς τεράστια ποσά εάν ε, γίνονται τέτοιου είδους ε, πολιτικές ε, αλλαγές. Δηλαδή, ανοίγουμε, κλείνουμε, ε, λέμε ναι, λέμε όχι. Από μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή, εντάξει, να αποφασίσουμε ότι το κλείνουμε, εντάξει, είναι μια απόφαση της χώρας. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορεί να αλλάξουμε ξανά, γιατί αλλιώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ε, κινητοποιήσουμε τις, τους απαραίτητους πόρους ε, για να προχωρήσουμε στην, ε, στις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξασφαλίσουμε την προμήθεια ενέργειας. Ένα ερώτημα ίσως ε, μπορώ να το θέσω κάπως διαφορετικά. Έχει αναφέρει η κυρία Σίζελη τη δική μου χώρα για το θέμα αυτό της επιλογής να μην ακολουθηθεί πυρηνική ενέργεια. Θα το εδιευρύνω το θέμα αυτό. Θα μπορούσε η πράξη της Γερμανίας να έχει μιμητές, ότι θα μπορούσαν και άλλες χώρες. Εσείς είπατε ότι δεν είναι ιδιαίτερα ε, πιθανό. Αλλά τι θα γινότανε στην πραγματικότητα αν στην Ευρώπη πολλά ή όλα τα κράτη ακολουθούσαν το παράδειγμα της Γερμανίας. Τι θα σήμαινε αυτό για την ασφάλεια εφοδιασμού ηλεκτρισμού, για το διοξείδιο του άνθρακος και για τις τιμές. Μήπως θα έπρεπε να συζητήσουμε αυτό το ερώτημα ποιες θα ήταν οι δυνητικές εξελίξεις αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πολύ ενδιαφέρον θέμα κύριε Πρόεδρε. Αν πολλές χώρες ακολουθούσαν την ε, απόφαση της Γερμανίας να υπάρξει σταδιακή εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας, η Ευρώπη το να χάσει λοιπόν την πυρηνική επιλογή σημαίνει, όπως <clears throat> θέλησα να δείξω, στην περίπτωση της Γερμανίας, η Ευρώπη θα, έχει, θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη εξάρτηση από τις ανανεώσιμες ενέργειες και οι ανανεώσιμες ενέργειες είναι πιο ε, πολυδάπανες και έχουν πολύ μεγαλύτερες διακοιμάνσεις. Επομένως χρειάζονται πολύ περισσότερες επενδύσεις για τα δίκτυα και για να υπάρχει και ε, υποστήριξη στην περίπτωση που δεν λειτουργούν <clears throat> οι αναλλακτικές ενέργειες θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη υποδομή φυσικού αερίου, όχι μονάχα σε ε, αέρια μορφή από τη Ρωσία αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Νότια Αφρική από τη Μέση Ανατολή. Αν όλη η Ευρώπη λοιπόν ακολουθήσει την γερμανική επιλογή αυτό θα σημαίνει σημαντική αύξηση εξάρτησης από ξένες πηγές φυσικού αερίου ή άνθρακος που θα δημιουργήσει μια τεράστια πρόκληση ενεργειακή ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη. Μπορείτε να το αποφύγετε, να το αποτρέψετε αυτό με αποφάσεις που θα λυθούν σε κάποια στιγμή. Γιατί αν γίνει η, απο, η αποχώρηση από την πυρηνική ενέργεια τόσο γρήγορα, οι ανανεώσιμες ενέργειες δεν μπορούν να καλύψουν το κενό τόσο γρήγορα. Λοιπόν, ενδιάμεσα υπάρχει ανάγκη να καλύψει κανείς το χάσμα. Η Γερμανία μπορεί να το κάνει γιατί οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να διαδρούν την πυρηνική ενέργεια. Επομένω, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, η Γερμανία μπορεί πάντα να βασιστεί στη γαλλική πυρηνική ενέργεια ή στην ε, ενέργεια που έρχεται από το κάρβουνο στην Πολωνία ή στην Τσεχία. Αν όλοι ακολουθήσουν την ίδια κατεύθυνση όμως της Γερμανίας, ο κίνδυνος να υπάρξουν κάποιες διαταραχές οι οποίες δεν μπορούν να απορροφηθούν αρκετά γρήγορα, εξακολουθεί να παραμένει. Πιστεύω λοιπόν ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, υπάρχει πολύ, πολύ μικρότερη ασφάλεια και μπορεί να προκύψει πολύ υψηλότερο κόστος ηλεκτρισμού και συγχρόνως ο άνθρακας είναι μια πολύ ελκυστική επιλογή αυτή τη στιγμή. Αυτό θα αυξήσει τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και για το λόγο αυτό πιστεύω η πρόκληση ενώπιον της οποίας βρίσκεται η Ευρώπη εάν θέλει να πετύχει τους στόχους του Κοπενχάγης τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακος, αυτό σημαίνει θα χάσει την ηγεσία που έχει η Ευρώπη για τη μείωση του διοξιδίου του άνθρακος σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Δεν υπάρχει κανένα άλλο ο οποίο θα αναλάβει τον λόγο. Ήταν πάρα πολλέ ερωτήσει Με ένα εκπληκτικό τρόπο έχετε απαντήσει κάθε φορά. Είμαστε ευγνώμονε γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν πράγματι μια αξιέπαινη ε, συζήτηση. Χαιρόμαστε που κάνατε αυτή την προσπάθεια να μπορούμε να κάνουμε αυτή την συζήτηση πριν από τις διακοπές. Ήταν εμπλουτιστική αυτή η συζήτηση για όλους Βέβαια πρέπει να λάβουμε μερικές σοβαρές αποφάσεις και είναι πάρα πολύ χρήσιμο που υπάρχουν αυτές οι πληροφορίες. Ξέρω ότι θα συναντήσετε την κυρία Μέρκελ την επόμενη εβδομάδα και θα της προτείνετε από ό,τι ξέρω, από ό,τι φαντάζομαι, να στείλει ένα γράμμα ευχαριστία σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίε κάνουν δυνατή τη γερμανική πολιτική. Λοιπόν, αυτό το λέω βέβαια υπομορφία θεϊσμού. αστεϊσμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Τανάκα. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε και ήταν πολύ θετικό που μπορέσαμε να συζητήσουμε μαζί μας. Σας ευχόμαστε κάθε τύχη. Okay, sind die anderen schon da? Okay, we can start, please, ladies and gentlemen, with the next point. Μπορούμε να ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο. Hello, welcome. Yeah.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 Συνεχίζουμε, εντάξει. Έχουμε χάσει λίγο χρόνο, αυτό είναι κακό, αλλά θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στο δυνατόν περισσότερο. Το επόμενο θέμα που έχουμε να εξετάσουμε προέκυψε από μια συζήτηση στην Επιτροπή μας, γιατί πολλοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι θα έπρεπε να ακούσουμε την άποψη του Κοινού Κέντρου Ερευνών, ΚΚΕΡ, για τα αποτελέσματα του καταστροφικού σεισμού και του τσουναμιού στην Ιαπωνία και εφόσον υπάρχει τόσο ενδιαφέρον εγώ περίμενα θα υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο μόλον τούτο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Νοέλ και τον κύριο Ντεσάντη από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και χωρίς ε, μακρηγορία θα σας δώσω αμέσω το λόγο. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα πείτε για τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Τζοβάνι Ντισάντι, είμαι ο επικεφαλής του Ινστιτούτου για την Ενέργεια του ΚΚΕΡ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Ινστιτούτο του, του οποίου προείσταμε τα τελευταία χρόνια έχει εμπλακεί στην ανάλυση της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας. Βρισκόμαστε στο Πέτεν στην Ολλανδία όπου υπάρχει ο μόνος ερευνητικό αντιδραστήρας ο οποίος ανήκει ακόμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι ο αντιδραστήρας υψηλής ροής νετρονίων. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η έρευνα στον πυρηνικό τομέα και γι' αυτό ο Γενικός Διευθυντής μου με έθεσε επικεφαλής της ε, ομάδος, ε, της ειδικής μονάδος στο Κοινό Κέντρο Ερευνών που ασχολείται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ε, κρίση της Φουκουσίμα. <clears throat> Η πρότασή μου είναι η εξή τώρα. Θα σπάσουμε την ε, παρουσίαση σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα το παρουσιάσει ο Μαρκ Νοέλ, ο οποίος είναι ο αρμόδιος για το project ε, καθαρισμού, clearing house μάλλον πώς λέγεται, της, το σχέδιο παρακολούθησης του, των εκτενωμένων στη Φουκουσίμα και μετά θα έρθω εγώ και θα σας ε, πω μερικά περισσότερα για το, τη συμβολή του Κοινού Κέντρου Ερευνών στα τεστ αντοχή, στα stress test που θα γίνουν τώρα στην Ευρώπη για τους ποινικούς σταθμούς. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στο Μαρκ για την τεχνική ε, παρουσίαση των τεκτενωμένων στην περίπτωση Φουκουσίμα. Μάρκ. Ευχαριστώ Τζοβάνι. Λέγομαι Μάρκ Νοέλ και είμαι υπεύθυνο για <clears throat> το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Clearing House, το κέντρο συλλογής πληροφοριών σε σχέση με τη Φουκουσίμα και θα δούμε τώρα τι ακριβώς έγινε στο σταθμό Daiichi Φουκουσίμα, ποιες ήταν οι συνέπειες σε επίπεδο ραδιενέργειας και ποια είναι και η εμπλοκή του Κοινού Κέντρου Ερευνών στα θέματα αυτά. Ξεκινήσουμε για το τι έγινε στις 11 Μαρτίου. Είχαμε σαν <clears throat> αρχή ένα πολύ ισχυρό σεισμό με επίκεντρο μέσα στη θάλασσα και σαν αποτέλεσμα αυτού του σεισμού έκλεισαν αυτόματα ορισμένες μονάδες του πυρηνικού σταθμού στο Φουκουσίμα Ντάιτσι και Νταϊνί και στο Τοκάι στο Τόκιο. Και στην Ολογκάβα επίσης. Ένα μία ώρα περίπου μετά από τον ε, ε σεισμό ήρθε ένα τσουνάμι και όπως θα δείτε στην παρουσίαση αυτό οδήγησε στα κυριότερα προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμού. Είναι επίση ενδιαφέρον να λάβετε υπόψη ότι υπήρξε ένας κύριος ε, σεισμός αλλά πολλοί μετασυσμοί μετά από αυτόν και ένας από τους μετασυσμού ήταν κλίμακο 7 ρίχτερ με επίκεντρο πολύ κοντά στο σταθμό Φουκουσιμαντάκη και οδήγησε και σε προβλήματα αυτό ο μετασυσμό, λοιπόν. Εδώ βλέπετε επομένως το, την ε, άποψη από τον αέρα του σταθμού. Έχει έξι σταθμούς, ε, σταθμούς ε, πυρηνικού ζέοντος ύδατος. Βασίζονται σε, μια, σε ένα σχέδιο της General Electric και θα έχουμε και μερικά περισσότερα ε, λεπτομεριακά στοιχεία για το θέμα αυτό. Αναφέρθηκα στο τσουνάμι που ήταν το κύριο πρόβλημα, γιατί ήταν πρόβλημα είχε δύο κύριους αντικτύπους. Ο πρώτος ήταν ότι υπήρξε πλημμύρισμα του σταθμού και ουσιαστικά ξεπέρασε την ικανότητα του συστήματος ε, άντλησης που φέρνει θαλασσινό είδωρ για να ψήξει κύρια στοιχεία του αντιδραστήρα. Χάθηκε λοιπόν η δυνατότητα ψήξης, αλλά επιπλέον η χώρη όπου βρίσκεται ο κύριος ε, σταθμός εφεδρικού εφεδρικής ισχύω με δίζελ, έχασε και αυτό την ικανότητα παραγωγής και εφεδρικής ισχύω. Βλέπετε λοιπόν την κατάσταση πριν και μετά από το τσουνάμι. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές δομές οι οποίες βρίσκονται κοντά στον όρμο που είναι η Φουκοσίμα που ουσιαστικά εξαφανίστηκαν. Βλέπετε παραγωγός ότι εδώ υπήρχαν ε, δεξαμενές οι οποίες εξαφανίστηκαν μετά από το τσουνάμι. Εδώ βλέπετε την έλευση του τσουναμίου στον πυρηνικό σταθμό βλέπετε ότι υπάρχει ένα τσιμεντένιο φράγμα το οποίο κανονικά θα έπρεπε να σταματήσει το τσουνάμι δεν έφτασε για να το κάνει αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλο το ύψος του τσουναμιού εδώ βλέπετε τώρα μια φωτογραφία μέσα στο σταθμό Αυτός ο, αυτή η αίθουσα είναι μεταξύ της αίθουσας που είναι οι στρόβιλοι οι στρόβιλογεννήτριες, οι τουρμπίνες και το, του πυρηνικού σταθμού αυτού καθεαυτού. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλο, μεγάλη ήταν η ένταση του τσουνάμι με τις καταστροφές που προξένησε σε αυτό το χώρο. Ναι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο, είναι εύγλωτες οι εικόνες. Λοιπόν, τώρα σας δείχνω την, το σχεδιασμό του πυρηνικού σταθμού γιατί είναι απαραίτητο να καταλάβετε την αλληλουχία των γεγονότων. Ο σταθμός του Φούκου Σιμαντάιτσι βασίζεται στο σχέδιο, General Electric Mark 1 είναι αντιδραστήρα ζέοντος ύδατος, δηλαδή ότι μέσα στον ε, αντιδραστήρα έχετε τον πυρήνα και έχετε είδωρ και επομένως μέσα στο κέλυφος αυτό έχετε ε, νερό το οποίο ψύχει τον ε, πυρήνα του αντιδραστήρα παράγεται ατμός ο οποίος πηγαίνει στις <clears throat> στροβιλογεννήτριες οι οποίες οδηγούν τους την παραγωγή ηλεκτρισμού και μετά το ατμός πηγαίνει σε ένα συμπυκνωτή, μετά πηγαίνει στο σύστημα ψήξη και ξαναγυρίζει στον πυρήνα του αντιδραστήρα. Ο πυρήνας βρίσκεται μέσα στο σύστημα, στο κέλυφος συγκράτησης το οποίο είναι μεταλλικό και έχει ένα παράξενο όπως βλέπετε σχήμα εδώ. Είναι αχλαδοειδής και έχει και δύο περαιτέρω θαλάμους ε, που θα επανέλθω σε αυτούς. Ας πούμε προς το παρόν ότι είναι ένα μεταλλικό κέλυφος. Λοιπόν, τι γίνεται. Ξεκινάει με το σταθμό η αλληλουχία των γεγονότων. Χάνεται η ηλεκτρική ισχύς. Εκείνη τη στιγμή οι αντιδραστήρες δεν έχουν υποστεί ζημίες. Υπάρχει η λεγόμενη διαδικασία Scrum, ότι αυτόματα κλείνουν οι αντιδραστήρες, αλλά όπως ξέρετε ακόμα και όταν κλείνει ένα αντιδραστήρες, υπάρχει ακόμα η υπολοιπόμενη ισχύση η οποία παράγεται από τον αντιδραστήρα, επομένω χρειάζεται ακόμα να υπάρξει ψήξη του αντιδραστήρα, ακόμα και μετά το σταμάτημα του αντιδραστήρα. Κανονικά ξεκινούν οι εφεδρικοί ε, diesel, και όλα δεν είναι καλό, αλλά περίπου μια ώρα αργότερα φτάνει το τσουνάμι στον πυρηνικό σταθμό, πλημμυρίζει την αίθουσα που είναι εφεδρική, ε, οι εφεδρικές γεννήτριες δίζελ και το αποτέλεσμα υπάρχει απώλεια ενέργειας ηλεκτρική σε σταθμό παραμένουν μονάχα οι εφεδρικοί συσσωρευτέ, οι μπαταρίες. Σε λίγο φυσικά οι μπαταρίε σταματούν να λειτουργούν γιατί έχουν εξαντληθεί και επομένω, από εκείνη τη στιγμή οι αντιδραστήρες 1 με 3 δεν έχουν κανένα τρόπο να απάγουν τη θερμότητα που παράγεται στον πυρηνικό σταθμό. Τι γίνεται αν δεν υπάρχει δυνατότητα απαγωγή θερμότητα. αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να δημιουργείται θερμότητα στον πυρήνα του αντιδραστήρα, έχετε όλο και περισσότερο ατμό ο οποίο παράγεται. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξετε τη βαλβίδα ασφαλείας γιατί αλλιώς θα υπάρξει υπερβολική πίεση στο κέλυφος. Όταν ανοίγεται όμω αυτή τη βαλβίδα ο, ο ατμός φεύγει στην ατμόσφαιρα και μειώνεται το επίπεδο του ύδατος στον πυρηνικό στον πυρήνα του εντραστήρα και αρχίζει να εκτίθεται στην ατμόσφαιρα ο πυρήνας. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η θερμοκρασία Υπάρχει ένα σημείο στους 1200 βαθμούς όπου η επένδυση των ε, ράβδων καυσίμου γύρω στους 1200 βαθμούς υφίστανται μια εξωθερμική αντίδραση μεταξύ του, του ζυρκονίου που βρίσκεται στους, ε, στην επένδυση και του ατμού που βρίσκεται στον θάλαμο πίεσης και αυτή η διαδικασία παράγει οξύδιο του ζυρκονίου και υδρογόνο. Στους σταθμούς 1 και 3 αυτή η συσσόρευση ο υδρογόνου που παράγεται από αυτή την αντίδραση και που συσσωρεύτηκε στο άνω μέρος του κελίφους οδήγησε σε μία έκρηξη και νομίζω τα έχετε δει αυτά με τα βίντεο στις, ε, στις ειδήσει. Εδώ βλέπετε το πάνω πάτωμα του αντιδραστήρα. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο, ε, μια μεγάλη πλάκα με ε, τσιμέντο που προστατεύει το σταθμό και απάνω έχετε τους σταθμούς όπου τίθενται τα ράβδη καυσίμου για να κρυώσουν και υπάρχει και το κέλφος το μεγαλύτερο το οποίο καλύπτει που, ε, προστατεύει τους, τα, του, τα εξαντλημένα καύσιμα του περιβάλλοντος. Και εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη ζημία από την έκρηξη υδρογόνου. Στην περίπτωση του, της μονάδος 2 η έκρηξη δεν έγινε στο πάνω μέρος αλλά στο κάτω μέρος και αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί εκεί πέρα υπήρξε απόλυτη διάρρηξη του κελίφου συγκράτησης και ανοίχθηκε προς την ατμόσφαιρα. Εδώ βλέπετε λοιπόν μετά από τις εκρήξεις υδρογόνου τον χώρο των πυρηνικών σταθμών. Σας είπα τι έγινε λοιπόν από τους ε, σταθμούς 1 και 3 και υπήρξε και μία έκρηξη στο σταθμό 4. Στην αρχή θεωρήθηκε ότι ήταν το αποτέλεσμα εκρήξεων στα πυρηνικά καύσιματα εξαντλημένα που βρισκόντουσαν στις δεξαμενές ψήξεις, αλλά είδαμε στη συνέχεια ότι δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο πιστεύουμε τώρα είναι ότι υπήρχε μια διασύνδεση των ε, σταθμών 3 και 4 και υπήρξε επομένω και συσσόρευση υδρογόνου. Βλέπετε εδώ πέρα ποια είναι η κατάσταση μετά από τις εκρήξεις υδρογόνου. Βλέπετε το, τις δεξαμενές ψήξεις για τα εξαντλημένα καύσιμα από που βγαίνει αυτή τη στιγμή ατμός, γιατί κάποια στιγμή υπήρξε υπερθέρμανση, γιατί δεν υπήρχε πια νερό στους, ε, στις δεξαμενές ε, ψήξεις. Υπήρξε ένα ρομπότ το οποίο εστάλει για να παρακολουθήσει την κατάσταση εκεί. Βλέπετε στο, στην μονάδα 4 ότι δεν υπάρχει μεγάλη καταστροφή, αλλά στη μονάδα 3 βλέπετε ότι υπήρχαν πολλά συντρίμια, ότι ουσιαστικά υπήρξε ένα μπάχαλο στο τμήμα, στο, στη μονάδα 3 και επομένως υπήρξε μεγάλη καταστροφή. Έρχομαι τώρα στις ε, ενέργειες αποκατάστασης για να μπορέσει να ε, περισταλεί η εξέλιξη του ατυχήματος. Βέβαια πολλές <clears throat> δράσεις είχαν σαν στόχο το να επανέλθει το ψυχτικό σύστημα. Άρχισε καταρχήν να υπάρχει ψεκασμός ύδατος κατευθείαν πάνω στις δεξαμενές ψήξεως και συνεχίστηκε και η, ε, η έγχυση θαλασσινού ύδατος προς τον, στο σύστημα ψήξης. Υπήρξε βέβαια ε, ε, διέρευσε ραδιενεργό νερό και έφτασε ως τη θάλασσα. Έγινε μια προσπάθεια να βρούμε τους τόπους όπου να βρεθούν οι τόποι από όπου γινόταν η διαρροή και να σταματήσουν με διάφορα φράγματα που εμπόδισαν την εκροή των νερών δημιουργήθηκε και ένα αρκετά ε, πλήρες πλαίσιο ε, εποπτείας της ραδιενέργειας που εκραίει στη θάλασσα και θα σας δώσω στοιχεία και γι' αυτό αργότερα. <clears throat> Περνάω τώρα αυτό εδώ πέρα, δεν σας λέω τίποτα για αυτό το θέμα, όπου ξέρετε ότι θα δημιουργηθεί ένα ε, προσωρινό κέλφος γύρω από τη μονάδα 1, το οποίο είναι υποκατασκευή. Εδώ σας δείχνω την τάση τάξη μεγέθους της ε, ε, συνολικής ραδιενεργής ε, δραστηριότητας που εκλήθηκε στο περιβάλλον. Το συγκρίνουμε για το, με το Τσερνομπίλ που είναι 5,2 εκατομμύρια τέρα μπεκερέλ. Στη Φουκουσίμα βρισκόμαστε σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο, περίπου 10 φορές λιγότερη συνολική ραδιενέργεια εκλήθηκε σε σχέση με το Τσερνομπίλ στην Φουκουσίμα. Εδώ βλέπετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η διαφάνεια γιατί δείχνει τις ε, μετρήσεις ακτινοβολίας γάμα σε διάφορα σημεία του πυρηνικού σταθμού. Βλέπετε ότι έχετε κορυφές δραστηριότητος που συνδέονται με τις ε, εκρήξεις που έγιναν ή με το γεγονός ότι άνοιξαν βαλβίδες ασφαλείας επίτηδες για να μειωθεί η πίεση του ατμού, αλλά μετά από το τέλος του Μαρτίου δεν υπάρχουν τέτοιες κορυφώσεις στην εκπομπή ε, ακτινοβολίας γάμα και βλέπετε την εκθετική μείωση της εκπομπής. Ε, ζώνες εκενώσεων τώρα, τι είναι για την προστασία του πληθυσμού. Ήδη την πρώτη μέρα, τη μέρα που έγινε ο και το τσουνάμι, υπήρξε εκένωση μια ζώνης τριών χιλιόμετρων γύρω από το πυρηνικό σταθμό την επόμενη μέρα, επειδή αυξήθηκε η πίεση μέσα στο κέλφος η, και επειδή ήταν γνωστό ότι θα πρέπει να υπάρξει έκκληση ατμού στην ατμόσφαιρα, <clears throat> αυξήθηκε η ακτίνα εκένωση στα 10 χιλιόμετρα. Την Κυριακή 13 έγινε η πρώτη έκρηξη στην μονάδα 1 και αυξήθηκε η εκένωση στους, στα 20 χιλιόμετρα. Αυτό σημαίνει ότι 170.000 κάτοικοι χρειάστηκε να να εκενωθούν. Δόθηκαν επίσης ταμπλέτες ιούδιου για να αποφευθούν προβλήματα στο θηροειδή. Υπήρξε έλεγχο στον πληθυσμό. Λοιπόν, μόνο 25 άτομα από το γενικό πληθυσμό φάνηκαν να έχουν μολυνθεί από ραδιενέργεια. 15 Μαρτίου αποφασίσανε να διευρύνουν τη ζώνη εκένωση στα 30 χιλιόμετρα και να απαγορευτεί η υπέρπτυση αεροπλάνων. Σιγά σιγά έγιναν μετρήσεις ε, σε διάφορα σημεία με αυτοκίνητα και με αεροπλάνα και εντοπίστηκε σημαντική ραδιενέργεια σε ένα νησί Μητατέ που είναι σε απόσταση 40 χιλιόμετρων έξω δηλαδή από, το, από την ζώνη ε, εκένωσης, το Ινιτάτε και βάσει αυτού αποφασίστηκε να υπάρξει επέκταση της ζώνης ε, εκένωσης που είναι τώρα τα 20 χιλιόμετρα και μια ιδιαίτερη περιοχή γύρω από αυτό το χωριό. Και θα εξηγήσουμε μετά γιατί είναι κάτι τέτοιο. Εδώ βλέπετε τώρα τις ε, <clears throat> επίγειες μετρήσεις. Βλέπετε ότι δεν είναι ομοιόμορφη η κατανομή της ραδιενέργειας, εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες, τη βροχή και το χιόνι μετά από τις ε, κρίξεις. Και βλέπετε ότι η ζώνη εκένωσης περιλαμβάνει και περιοχέ όπου ανέμενε ο πληθυσμό ένα χρόνο θα έπαιρνε μια συνολική δόση 20 μιλισίβερ μέσα το γρό. Το χρόνο δεν είναι τεράστια αυτή η ποσότητα, είναι αρκετά συντηρητική αυτή η προφύλαξη που λαμβάνεται. Έχω τώρα να σας δείξω μερικέ ε, ε, διαφάνειες για να δείτε το πρόγραμμα ε, ραδιοεποπτείας. Ε, υπάρχουν ε, δείγματα τροφίμων που ελήφθησαν και δείχνει απλώς τον αριθμό των ελέγχων που έγιναν για τρόφιμα. Υπήρξαν πολλά θετικά, θετικές μετρήσεις που ξεπερνούσαν τις τιμές ασφαλείας και βλέπετε σε ποιους τόπους έγιναν αυτά. Υπήρξαν πιο λεπτομερείς απαγορεύσεις ορισμένων προϊόντων. γιατί υπήρξε ραδιενέργεια πάνω από το όριο το οποίο επιτρέπεται για πολλά λαχανικά, για γάλα, για ψαρία κτλ η ασφάλεια του πόσιμου ύδατος. Υπήρξαν ορισμένε απαγορεύσει σε ορισμένες επαρχίε. Αν δούμε το Τόκιο, υπήρξε απαγόρευση μόνο για τα βρέφη και μόνο για μία μέρα. Μετά οι μετρήσεις ήταν πάντα κάτω από το όριο ασφαλείας για τους ενήλικες. Και τέλος, υπήρξε μεγάλη καταμέτρηση ραδιενέργειας στη θάλασσα και βλέπετε εδώ για το Κέσιο 137 ότι ήταν και χρήσιμες αυτές οι μετρήσεις για να εντοπιστεί η πηγή διαρροής ραδιενεργών υδάτων και από τη στιγμή που έγινε αυτός ο εντοπισμός βλέπετε την ε, βαθμία μείωση της ε, δραστηριότητας της ραδιενέργειας στο, στα ύδατα της θάλασσας. Και δίνω τώρα το λόγο στο, στον κύριο Ντεζοβάνη, Ντεσάντι. Περνάμε στο δεύτερο κομμάτι τώρα της παρουσίασης για να καταλάβουμε πόσο το GRC μπορεί να βοηθήσει και να επικουρήσει την Επιτροπή της Κομισιόν την Task Force. Η Task Force δημιουργήθηκε από τον πρόεδρο Μπαρόζο και θέλει καταρχάς να επιβλέψει την εφαρμογή των stress test και να υποβάλει μια πρώτη, ένα πρώτο σχέδιο έκθεσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο 2011 και δεύτερον να αναλύσει τα μέτρα προστασίας από τη ραδιενέργεια τα οποία συζητήθηκαν στην Ευρώπη και να προτείνει ε, διορθωτικές ενέργειες. Ε, ούτως ή άλλως η ενακτήρια συνεδρίαση έγινε τον Ιούνιο φέτος. Μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου όλες οι εκθέσεις πρόοδου από τους εθνικούς ρυθμιστές θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτως ή άλλως πολλοί έχουν κάνει μια αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας θα υποβάλουν ε, τα σχέδια στους εθνικούς, ε, στις εθνικές αρχές και μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα σταλούν τα προκαταρκτικά εθνικά, ε, εθνικές εκθέσεις. Μέχρι μέσα Νοεμβρίου επομένως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συντάξουμε, να συντάξουμε το πρώτο σχέδιο της έκθεσης για να είμαστε έτοιμοι ε, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Όμως την ανάλυση των εκθέσεων θα τη συνεχίσουμε και ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε και τις, ε, τις τελικές εθνικές εκθέσεις. Μέχρι το, στις 30 Απριλίου του 2012 θα ολοκληρωθεί η peer review και ε, θα είμαστε έτοιμοι επομένως για να υποβάλουμε την τελική ανάλυση και την τελική έκθεση τον Ιούνιο του 2012. Τώρα, το GRC, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, είμαστε, είναι το μόνο που μπορεί να κάνει άμεση έρευνα. Γι' αυτό θα, θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την task force. Γιατί εμείς έχουμε την εμπειρία στα θέματα πυρηνικής ασφάλειας. Και εδώ και δύο χρόνια επίσης έχουμε δημιουργήσει αυτό το περίφημο European House. Experience Project είναι ένα project το οποίο μας το ζήτησαν πολλές αρχές ασφάλειας κρατών μελών γιατί ήθελαν να δι... δημιουργηθούν ε, αρμοδιότητες στα θέματα πυρηνικής ασφάλειας γι' αυτό ήθελαν να ε, εποφεληθούν από τα διδάγματα και από τις εμπειρίες και από τις πρακτικές που εφαρμόζαν οι χώρες που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια εδώ και καιρό. Επομένως εμείς συντονίζουμε, αν θέλετε, συγκεντρώνουμε όλα αυτά τα ε, στοιχεία και όταν έγινε το επεισόδιο στην Φουκοσίμα μπορούσαμε να ε, μοιράσουμε τα στοιχεία αυτά που σας παρουσίασε ο Μάρκα σε όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι στιγμής όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν, ε, συμμετέχουν σε αυτό το clearing house ε, project. Τώρα βέβαια θα πρέπει να προχωρήσουμε ε, και στην ανάλυση των όλων των συμβάντων στη Φουκοσίμα. Αυτή είναι η οργάνωσή μας, το βλέπετε, ότι αριστερά έχουμε τα κράτη του Clearing House, που είναι τα πλήρη μέλη και του παρατηρητές, Όλα τα κράτη-μέλη βρίσκονται εδώ. Και υπάρχει και μία επιτροπή, ε, συντονιστική επιτροπή, η οποία ε, συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και ε, υποβάλλουμε ένα, μια έκθεση και στην, στο Διεθνή Οργανισμό Πυρηνικής Ενέργειας στη Βιέννη και στο ΝΙΑ, στο, στο Clearing House όλα αυτά, αυτό το project ήταν και χρήσιμο και πριν τη Φουκοσίμα. Τώρα είμαστε ακόμα πιο χρήσιμοι, ακόμα πιο χρήσιμο και πολύτιμο. Διότι γινόμαστε ένα ευρωπαϊκό κλάμπ εμπειρογνωμόνων, εάν θέλετε, και καταλήγουμε σε κάποια, κάνουμε κάποια ανάλυση, σε κάποια συμπεράσματα κτλ. Αυτό μας επέτρεψε να Εδώ και αρκετό χρόνο εμείς έχουμε την, τις γνώσεις που απαιτούνται και προσφέρουμε τεχνική υποστήριξη στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Ε, ξέρουμε τους διαφορετικούς τύπους των πυρηνικών αντιδραστήρων, ακόμα και των παλαιών που είχαμε στο παρελθόν στην Ευρώπη. Και συνεργαζόμαστε ε, και με όλες τις ε, αρχές πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Clearing House. Και με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε, αν θέλετε, μια κοινή δεξαμενή, αν θέλετε, ε, γνώσης. Και μπορούμε να προσφέρουμε και δυνατότητες συνεργασίας και με γειτονικές χώρες πρακτικά πλέον στην γίνεται. Μέχρι στιγμής τι κάνουμε. Κάθε μέρα συγκεντρώνουμε στοιχεία από τους Ιάπωνες συναδέλφους και τα διανύμουμε τα στοιχεία αυτά στους συναδέλφους του Clearing House, δηλαδή λίγο πολύ σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά ε, έχουμε συνεισφέρει στην, ε, στον ορισμό του στόχου και στη μεθοδολογία για, τα, για τις δοκιμασίες ε, και θα συνεισφέρουμε ούτως ή άλλως στον ορισμό των κοινών κριτηρίων. Την επόμενη Δευτέρα θα συζητηθούν τα θέματα αυτά στην ε, Κομισιό. Επομένως, θα, ορίσουμε ε, για το, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και πώς θα γίνει η συμμετοχή μας σε διάφορα task force και σε συνεργασία με τους ρυθμιστές και μετά όπως σας είπα όταν ε, έχουμε διαθέσιμες τις εθνικές αναφορές θα προετοιμάσουμε την αναφορά για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επίσης θα υποστηρίξουμε οποιαδήποτε διεθνή δραστηριότητα όσον αφορά την ανάλυση των κινδύνων εφόσον υπάρχουν χώρες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας και να το κάνουμε από κοινού. Επομένως, προσπαθούμε να συνδυάσουμε την επιστημονική πτυχή των ε, stress test. Ε, συζητάμε ακόμα βέβαια με τις διάφορες χώρες τι θα γίνει και πώς θα γίνουν όλα αυτά, αλλά για την Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η, γενική, η συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση ε, θα συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Αυτά ήθελα να πω ε, εν συντομία και πολύ συγκεκριμένα και αυτά θα, αυτά θα γίνουν, ε, δηλαδή για να σας πω ποια θα, θα είναι η δραστηριότητά μας στις επόμενους μήνες. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεσάντη για τις πληροφορίες που μας δώσατε και ξέρουμε τώρα τι ακριβώς μπορούμε να περιμένουμε για το μέλλον. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά να τα ξέρουμε. Κυρία Σίζελ, έχετε το λόγο και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Θέλω να σας ρωτήσω για τη διαδικασία όσον αφορά τα τεστ αντοχής. Η διαδικασία αυτή πάει πολύ γρήγορα, είναι πολύ συγκεκριμένη και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ως εμπειρογνώμονες που είσαστε, τι αποτελέσματα περιμένουμε και τι συνέπειες θα υπάρχουν τη στιγμή που λίγες εβδομάδες έχουν οι αρμόδιοι στα κράτη-μέλη ρυθμίσεις. Αυτή η διαδικασία λοιπόν είναι δυνατόν να είναι τόσο γρήγορη και τόσο σύντομη όταν πρόκειται για ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Ίσως μπορείτε να απαντήσετε άμεσα, αν θέλετε. Ευχαριστώ για την ερώτηση που δεν είναι βέβαια και εύκολη ερώτηση γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, δύο διαφορετικές ανάγκες. Απ' τη μια θέλουμε μια σε βάθο ανάλυση όλων των πτυχών, απ' την άλλη βέβαια πιέζει ο χρόνος. Το Συμβούλιο, οι πολίτες περιμένουν πολύ γρήγορα να έχουν αξιόπιστα αποτελέσματα. Εμείς αναμένουμε να έχουμε μια πλήρη ανάλυση όσον αφορά την ασφάλεια των αντιδραστήρων και να συμπεριλάβουμε και εξωτερικά συμβάντα, πράγματα τα οποία κάθε φορά αναλύονται και επαναξιολογούνται. Προσπαθούμε όμως όσο γίνεται πιο γρήγορα να εφαρμόσουμε τα κριτήρια αξιοπιστίας που έχουμε. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε συμπεράσματα για να δούμε τι μπορούμε παραπέρα να κάνουμε. Πιστεύουμε πάντως ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να κάνουμε αυτή την αξιολόγηση. Αλλιώς χρειάζονται χρόνια αν θέλετε να έχουμε μια πραγματικά πλήρη και σε βάθος ανάλυση όλων των πτυχών. Έπειτα υπάρχει το θέμα των αδειών, υπάρχει το θέμα των, ασφα... αρχών ασφάλειας, υπάρχει και το θέμα της διαδικασίας. Το θέμα είναι να είμαστε αξιόπιστοι απέναντι στον Ευρωπαίο πολίτη ώστε να υπάρχει μια εναρμονισμένη προσέγγιση με διαφάνεια και επιστημονικά ορθή. Πιστεύω ότι όντως αυτό είναι το πιο δύσκολο και μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Η Ευχαριστώ. Πόσο συνεπή είναι τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή των, ε, δοκιμασιών αντοχής έχω ακούσει τον κύριο Βάιτμαν στην Πολυ... στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, που αναφέρθηκαν, ε, αναφέρεται στην, αναφέρθηκε στην έκθεση η οποία συντάχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, το, η οποία όμως δεν αναφέρθηκε στα προηγούμενα ε, τεστ, stress test. Θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη καλύπτουν όλους τους ε, τομείς ε, που εσείς ε, και η Επιτροπή έχει καθορίσει, έχετε καθορίσει και τι διαδικασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν κάνετε την peer review, να φτάσετε σε εκείνο το στάδιο, τι μπορείτε να κάνετε εάν βρείτε ότι τα κράτη-μέλη δεν ήταν τόσο ενδελεχή και συνεπή στην ανάλυση που κάνανε. Ε, έχετε κάποια, κάποιο τρόπο να επιμείνετε και να πείσετε τα κρατημέλη να κάνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Για τον απλούς λόγο ότι η άσκηση αυτή θα γίνει από κοινού με τις εθνικές αρχές ασφάλειας. Δηλαδή έχουν οι, αρμόδιε οι αρμόδιες αρχές έχουν την ε, δυνατότητα, έχουν την εμπειρογνωμοσύνη να το κάνουν. Όπως σας είπα και προηγουμένως, συζητάμε ακόμα με τις ε, αρχές ασφαλείας και θα, η, τελική εκδοχή της μεθοδολογίας ε, για τα stress test θα ε, δημοσιευθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε και να αναλύσουμε όλες τις εκθέσεις που έχουμε πάρει και μετά να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, διότι υπάρχουν εθνικές εκθέσεις μεν, αλλά χρειαζόμαστε και μία ομοιογένεια. Ε, υπάρχουν τρεις διαφορετικές ομάδες ε, που οριζόντια αναφέρονται σε τρία διαφορετικά θέματα, εξωτερική κίνδυνη, σοβαρά ατυχήματα και ένας άλλος τομέας και μετά θα πρέπει να δούμε πώς κάθε εθνική έκθεση απαντά σε αυτούς τους τρεις ε, διαφορετικούς τομείς. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε πώς οι εκθέσεις αυτές ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουμε προτείνει. Γι' αυτό ξοδεύουμε και τόσο χρόνο για να καθορίσουμε τις παραμέτρους, τα κριτήρια, τις προσδοκίες μας από τις διάφορες εθνικές εκθέσεις. Και θα είμαστε αυστηροί ε, όταν κρίνουμε τις εκθέσεις. Θα εντοπίσουμε τα κενά και θα ζητήσουμε να καλυφθούν. Γιατί στο κάτω-κάτω θα, θα αμφισβητηθεί και η αξιοπιστία αυτής του όλου εγχειρήματο. αν δεν γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει. γιατί οι πληροφορίες ε, στα μέσα ενημέρωσης ίσως ήταν διωγγωμένες και δραματοποιημένες. Ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι ακριβώς είχε γίνει και να καταλάβει ποια ήταν τεχνικά έγκυρα και ποια όχι. Εγώ θέλω να θέσω το ερώτημα. Σε σχέση με το πρόβλημα αυτό, στη Φουκουσίμα σε ποιο βαθμό ήταν κάτι το οποίο έγινε λόγω της βίαιης δράσης της φύσης ή αν οφειλόταν και στις τεχνικές ε, εγκαταστάσεις, τη μορφή που είχαν τεχνικές εγκαταστάσεις. Υπήρξαν, όπως είπατε, κάποιοι, υπήρξαν κάποιες καταγραφές σε βίντεο της καταστροφής και πολλές φορές ήταν πολύ χρήσιμες. Υπάρχει κάποια δυνατότητα να επεξεργαστεί κανείς αυτό το στοιχείο. Εγώ δεν έχω δει να έχει γίνει μια πρακτική αξιολόγηση. Μονάχα νέα, μονάχα πληροφορίες υπήρξαν. Αν ήταν, παραδείγματος χάρη, το προστατευτικό τείχος πιο ψηλό, θα είχε αποφευχθεί αυτό το ατύχημα. Επίσης, σε σχέση με τα μέτρα και τα, τις ενέργειες που έγιναν μετά από την καταστροφή, ήταν λανθασμένες οι ενέργειες που έγιναν και συνέτειναν στην ε, κατάσταση που δημιουργήθηκε ή όχι. Και σε σχέση με την καταστροφή στο Τσερνομπίλ, εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Όταν εμείς συζητήσαμε το θέμα αυτό στην ε, <clears throat> Ολομέλεια του Κοινοβουλίου όλα, όλες οι παρουσιάσεις είχαν ένα δραματικό χαρακτήρα αλλά θα θέλαμε να έχουμε και μία πιο συγκεκριμένη γνώση για το τι έγινε σε επίπεδο διάσωσης, ε, σε επίπεδο αποκατάστασης και θα ήθελα να ξέρω και πόσα άτομα τελικά έχουν ε, τραυματιστεί ή έχουν υποστεί προβλήματα από την ραδιενέργεια, οτιδήποτε. Ευχαριστώ. Πολλές οι ερωτήσεις σας. Πρώτον, το θέμα των ε, αξιόπιστων πληροφοριών που διατέθηκαν από την ε, Ιαπωνία μετά το ατύχημα. Οι Ιαπωνικές αρχές δημοσίευσαν ε, έκθεση σε επίπεδο IEA με διάφορα στοιχεία και λεπτομερείς πληροφορίες. Αν διαβάσετε την έκθεση αυτή θα καταλάβετε τι έγινε τις πρώτες μέρες με τα control rooms, τι μέσα είχαν στη διάθεσή τους που δεν είχαν ουσιαστικά. Έτσι κι αλλιώς ε, στους χώρους ε, επικρατούσε σκοτάδι, δεν ήταν εύκολο να κάνουν καμία διάγνωση της κατάστασης. Αυτό ήταν και ο κύριος λόγος για το ότι δεν είχαμε αρκετές πληροφορίες στη διάθεσή μας στην αρχή. Έπειτα, αναφερθήκατε στο τείχος που προστατεύει από το τσουνάμι. Αυτό το αναγνωρίσαμε. Υπήρξε και ερευνητική αποστολή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας και τα συμπεράσματα της ομάδας που πήγε εκεί ήταν ότι δεν είχε εκτιμηθεί όπως θα έπρεπε ο ενδυνάμει κίνδυνος. Είχε υποεκτιμηθεί. Αυτό είναι ένα από τα ε, μαθήματα που δυστυχώς πήραμε από αυτή την υπόθεση. Για την ε, ακτινοβολία τώρα. Πέρα από την ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα που υπήρξε και διαφορετικός τρόπος σε σχέση με το Τσερνομπίλ. Στο Τσερνομπίλ έγινε μια έκρηξη και διάφορα σωματίδια πήγαν σε ιδιαίτερα μεγάλο ύψος της ατμόσφαιρας. Ήταν διαφορετικό εκεί το φαινόμενο από ότι εδώ που εδώ υπήρχε διάχυση μέσα σε μια πιο μεγάλη χρονική περίοδο προς τη θάλασσα ως επιτοπλίστων ευτυχώς, και μέρος της ακτινοβολίας ε, πήγε στη θάλασσα. Άρα οι άμεσες επιπτώσεις πάνω στον πληθυσμό είναι διαφορετικές. Αυτά νομίζω με ρωτήσατε. Ευχαριστώ. Να προσθέσω και κάτι ακόμα η επιστημονική κοινότητα θα περάσει καιρός για να καταλήξει σε τελικά συμπεράσματα. Θα χρειαστούν χρόνια για να καταλάβουμε ακριβώς τι έγινε και να πάρουμε τα μαθήματα που πρέπει από το συμβάν. Ξέρετε ότι έτσι κι υπάρχει ένα νέο πρόγραμμα ε, κατάρτισης μετά από τόσα έγιναν στη Φουκουσίμα γιατί θα πρέπει με διαφάνεια να γίνει ανάλυση, να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε ώστε να αποφύγουμε κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Θέλουμε λοιπόν να ενημερώσουμε τους φοιτητές που ασχολούνται με τέτοια θέματα και γενικότερα τον πληθυσμό. Ήδη λοιπόν έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, είναι ευπρόσδεκτη και θα αποφασιστεί ποιο θα είναι ακριβώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που χρειάζεται και το οποίο θα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε. ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ίσως εάν χρειάζεται περισσότερη πληροφόρηση έχει να κάνει με αυτό που ανέφερε και ο Σδοβνόφσκι ότι χρειάζεται ίσως περισσότερη γνώση, περισσότερη ικανότητα ανάλυσης και καλύτερη συνειδητοποίηση των διαφορών μεταξύ του Τσενομπίλ και της Φουκουσίμα. Όλα αυτά σίγουρα μας βοηθούν στην αποδραματοποίηση, αλλά το ερώτημα είναι αν η Φουκουσίμα συμμορφωνόταν με τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί η Ευρώπη για τους πυρηνικούς σταθμούς. Αυτό νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον το ερώτημα. Χρησιμοποιήθηκε λαθασμένη τεχνική, ε, τι ακριβώς συνέβη. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι νομίζω το μοναδικό <clears throat> ουσιαστικό ερώτημα. Αν οι, τεχνο, οι, αν οι τεχνολογικές γνώσεις της εποχής εφαρμόστηκαν, αν χτίστηκε ο σταθμός και το περιβάλλον του με τον τρόπο που ανταποκρινόταν σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα, είναι ένα πράγμα να έχετε ένα κίνδυνο ο οποίο είναι απόλυτα απρόσμενο και δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και αν από την άλλη μεριά υπήρχε ένα κίνδυνο ο οποίο μπορούσε να ποσοτικοποιηθεί και να είναι γνωστό εκ των ε, προτέρων. Όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία και αυτό είναι το βασικό δίλημα το οποίο κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διευκρινίσει τη συζήτηση. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι μπορούμε να πούμε για το αν οι προδιαγραφές ήταν τέτοιες ώστε να μπορούσε να αποτραπεί το ατύχημα αυτό. Ναι, από επιστημονική άποψη όλα αυτά είναι αρκετά πρόωρα γιατί δεν έχουμε ακόμα τις πληροφορίες που χρειάζεται. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε όλα αυτά τα τεστ, αλλά σίγουρα θα υπάρξει μια μακρά επιστημονική διαδικασία για να αναλύσει τις συνέπειες, τα μαθήματα που διδαχτήκαμε από την καταστροφή, τα μέτρα ασφαλείας που μπορούν να βελτιωθούν. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ψηλό το επίπεδο ασφαλείας των ευρωπαϊκών πυρηνικών σταθμών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να σας δώσω μια απάντηση για το αν είναι ασφαλής η ευρωπαϊκή πυρηνική σταθμή, αλλιώς δεν θα χρειαζόμασταν καθόλου τα τεστ αντοχής. Αν δείτε τι έγινε μετά από το Three Mile Island και το Τσερνόμπιλ, χρειάστηκαν <clears throat> χρόνια μελετών για να καταλάβουν γιατί το σενάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε εκεί δεν το είχε προβλέψει κανείς εκ των προτέρων και υπήρξαν πάντα νέα στοιχεία ασφάλειας τα οποία έγιναν κατανοητά μετά. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και μετά από τη Φουκουσίμα και όλα αυτά που έχουμε κάνει είναι απλώς το πρώτο βήμα. Οπότε θα έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα, ξέρω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κάνουν προσπάθειες καλύτερης γνώσης και κατανόησης και ίσως κάποια μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν <clears throat> αμέσως. Αλλά τώρα σας πω, από τώρα πια αυτά τα μέτρα δεν θα ήταν σωστό, είναι πολύ πρόωρο. Θα υπάρξει και μία αξιολόγηση στα stress test. Θα υπάρξει μια, κατα... μια ε, κατανομή και μια αξιολόγηση για κάθε χώρα ξεχωριστά ή όχι. Ναι, θα πάρουμε την εθνική έκθεση από τις Εθνικές Αρχές Ασφαλείας θα τις ε, συνενώσουμε όλες, θα προσπαθήσουμε να τις δούμε οριζόντια, θα προσπαθήσουμε να δούμε αν απαντούν σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα με τον ίδιο τρόπο όλες οι εθνικές αρχές, να εξασφαλίσουμε αυτήν την ομοιογένεια και να εξασφαλίσουμε ότι η ποινική σταθμή είναι ασφαλή σε σχέση με το ΑΕΒ θέμα, αλλά θα κοιτάξουμε και την εθνική διάσταση θα έχουμε ουσιαστικά ένα πίνακα που να περιλαμβάνει και τα εθνικά στοιχεία. Θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, ομοιογένεια. Είναι καλό να ξέρει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι ό,τι και να συμβεί το επίπεδο ασφαλείας είναι το ίδιο. Αλλά να καταλάβουμε και σε επίπεδο κάθε κράτους τι δράσεις θα πρέπει να εφαρμόσουν και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Εντάξει. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι όταν έχετε τα στοιχεία αυτά είτε από εσά είτε από άλλου φορεί σε σχέση με τι πραγματικέ αιτίε τη καταστροφή Φουκουσίμα. Θα μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία. Και δεύτερον, είναι θετικό ότι η Ευρώπη απήντησε τόσο γρήγορα με τα τεστ αντοχής και ίσως αν μπορέσουμε να έχουμε ε, μεγαλύτερη να δούμε τα θέματα αυτά με μεγαλύτερη γαλήνη. Αυτό θα είναι κάτι που θα βοηθήσει πάρα πολύ την Ευρώπη όταν είναι σε δύσκολες στιγμές, ότι μπορούμε στην Ευρώπη να έχουμε κοινή δράση. Αυτό είναι ένα επιχείρημα που δείχνει πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή συνεργασία. Βρισκόμαστε σε εποχές που τέτοια επιχειρήματα υπέρ της ευρωπαϊκής συνεργασίας να είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τον κύριο Ντεσάντη και τον κύριο Νοέλ και όλους τους συναδέλφους Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή επένδυση χρόνου να ακούσουμε τις απόψεις και να πάρουμε πληροφορίες από εσά και έτσι μπορούμε... Α, κύριε Κορέα Δεκάμπος, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, σήκωσα και πριν το χέρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ τους εκπροσώπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Νιώθω ότι ήταν ένα προνόμιο να μπορέσω να έχω αυτά τα στοιχεία που έχω πάρει από εσά. Έχω παρακολουθήσει αντίστοιχε παρουσιάσει τη ΣΤΟΑ και ήταν πολύ θετικά αυτά που μα παρουσιάσατε. Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονό ότι έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλέ πληροφορίε, ενώ <clears throat> μόνο τρει μήνε ουσιαστικά έχουν περάσει από το ατύχημα και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει με εντυπωσιάζουν. Παραμένει για μένα μια τεχνική απορία ενός αδαούς. Τι έγινε με την χρήση θαλασσινού ύδατος για την ψήξη των αντιδραστήρων. Εγώ φαντάζομαι ότι ακόμα διοχετεύεται ε, θαλασσινό είδωρ για την ψήξη των αντιδραστήρων και αυτό το νερό στη συνέχεια περνάει σε ελεγχόμενες περιοχές. Από ό,τι είπατε, δεν υπήρξε ε, διαρροή αυτού του ύδατος. Ποια είναι τα τελευταία στοιχεία για την ραδιενέργεια στον ωκεανό, εάν έχετε τέτοια στοιχεία για, την, ε, <clears throat> το επίπεδο ραδιενέργειας στη θάλασσα. Ευχαριστώ. Δοθήκετε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ναι, η ψήξη του αντιδραστήρα γίνεται χρησιμοποιώντας ε, νερό και μετά από το περίβλημα βγαίνει και συσσωρεύεται στο χαμηλό τμήμα του αντιδραστήρα. Είναι δηλαδή ραδιενεργό είδωρ. Οι ανησυχίες για το ότι το νερό αυτό πάει στη θάλασσα, πρέπει να ξέρετε ότι εδώ ε, φροντίζουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να έχουν ε, ε, μηχανισμούς επεξεργασίας του νερού αυτού ώστε να καθαρίζει. και φροντίζουν να υπάρξει και αρκετός χώρος αποθήκευσης ώστε προσωρινά να μπορούν να κρατήσουν εκεί το ραδιενεργό είδωρο. Αυτή είναι η λύση προς το παρόν. Δεν έχω πια άλλη ερώτηση. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους. Σας εύχομαι ένα ήρεμο απόγευμα και μερσή και πάλι.